Αγαπητοί συναδελφοί, προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Λοιπόν, έχουμε εργαστεί πολύ πιο γλίγορα όποτε προβλέπετε από αυτές τα απόγευμα μέχρι τώρα και γι' αυτό έχουμε μόνο τρία θέματα ακόμα στη μεσαία διάταξή μας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προχωρήσουμε γρήγορα για να μπορέσουμε το γρηγορότερο δυνατόν να είμαστε ελεύθεροι, έχοντας εξετάσει βεβαίως βάθος τα θέματα που απομένουν. Έχουμε την έκθεση γνωμοδότησης του συναδέλφου Αλφόνση για τη Συμφωνία Αλίας με τις ε, νήσους του Προσύνου Προτερίου. Κατόπιν έχουμε τη ακρόαση του Αντιπροέδρου της ε, Σερβικής Κυβέρνησης και μετά έχουμε μία ψηφοφορία για την κινητοποίηση του τομείου Λεγγύης ε, για την ε, ε, παγκοσμιοποίηση της Βάρβαρα Μαρτέρα. Λοιπόν, ο Σέρβος Αντιπρόεδρος θα πρέπει να έρθει κανονικά στις 4 παρατέταρτο. Αν δεν είναι, για να μην χάσουμε καιρό, θα ζητήσω να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ορισμένοι συνάδελφοί μου είπαν ότι θέλουν οπωσδήποτε να είναι παρόντες για την ψηφοφορία, αλλά δεν θα μπορούν να έρθουν πριν από τα τέλη της, ε, του γιατί θα είναι σε μια άλλη επιτροπή. Τι να γίνει, θα αναγκαστώ να κάνουμε την ψηφοφορία γιατί δεν υπάρχει κύρια νομίζω διαφορά απόψε μεταξύ των πολιτικών ομάδων για αυτό το θέμα. Οπότε, εάν έρθει εγκαίρος ο Σέρβος Αντιπρόεδρος θα περάσουμε στην ακρόασή του πριν την ψηφοφορία, ε, αλλιώς θα ψηφίσουμε πριν για να κερδίσουμε χρόνο. Ωραία ο κύριος Φρανσουά Αλφονσί που να πάρει το λόγο και θα τον ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον για την ελευτική σύμπραξη ΕΕ Πρασινού Κριτηρίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξετάζουμε λοιπόν μία έκθεση για την Αλληλευτική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρασίνου Ακροτηρίου βάσει της νέας συμφωνία, συνθήκης της, Ρώμη, ε, Λισαβόνα. Συγγνώμη. Η πέμπτη Αλληλευτική Συμφωνία είναι που εξετάζουμε η πρόεδρος είναι η Σαλομονίδη Κομοράν, Σεϊχέλες και η Σαντομέ και Πριντσίπε. Η πέμπτη εδώ αφορά λιγότερο από 1,5 εκατομμύρια ευρώ το έτος. Για τρία χρόνια. 1,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή συνολικά. Από τις πέντε συμφωνίες ε, η πρώτη που ζητά ε, η γνώμη μας μέσα στις σωστές προθεσμίες μέχρι την πρώτη πρώτου του επόμενου έτος. Ε, μέχρι τώρα τα κάναμε με μεγάλη καθυστέρηση, τώρα όμως είμαστε στο χρονοδιάγραμμα. Δεν έχω πολλά να πω, είναι μια έκθεση στην οποία θα έλεγα να ψηφίσουμε θετικά. Θα ήθελα βέβαια να υπάρχει μια γενική μελέτη για τις συμφωνίες αυτής αλίας γιατί οι επόμενες θα έχουν σημαντικότερες δημοσιονομικές επιπτώσεις, μια δεκάδα εκατομμύρια ευρώ και θα ήθελα να μπορέσουμε και η δική μας Επιτροπή και η Επιτροπή Αλίας από κοινού να μελετήσουν αυτές τις συμφωνίες Αλίας με τις τρίτες χώρες. Πρόεδρος, θαυμάσια. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Η κυρία Ρελή. Απλώ ήθελα να υποστηρίσω το έτοιμο του κ. Αλφονσίν. Πολλέ φορές ε, είχαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνεδρίαση τη Επιτροπή και τη δική μα. Αν μπορείτε να το οργανώσετε στις κατάλληλε ε, προθεσμίες κ. Πρόεδρε. Γιατί προσεχώ θα έχουμε πραγματικά σημαντικές δημοσιογραφικές επιπτώσει για τι ε, δημιουργίε αυτέ τη μια κοινή συνάντηση των Επιτροπών Αλίας και Προπολισμού. θα ήταν σημαντική. Στηρίζω λοιπόν το έτοιμο του κ. Αλφονσί επί του θέματος. Πρώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, θεωρώ ότι πρόκειται για θέματα πάρα πολύ σημαντικά, ότι αυτές οι συμφωνίες συμπεριλαμβάνουν ενισχύσεις σημαντικές για την ανάπτυξη των εν λόγω δικαιούχων περιοχών ή χωρών Δεν ξέρω αν θα γνωμοδοτήσει και η Επιτροπή ανάπτυξη για αυτού του είδου τη ε, αλλά οπωσδήποτε έχουν κάποιο ενδιαφέρον για αυτήν. Και, όπω είπαμε, πρέπει να το κάνουμε επιτέλου, θα πρέπει να οργανώσουμε μια κοινή συνεδρία εργασία μεταξύ εκείνων τη Επιτροπής και προπολογισμών ίσω και ανάπτυξη για να καταλήξουμε σε μια κοινή στρατηγική. Μου φαίνεται σημαντικό. Η κυρία Ντουιρό έχει το λόγο. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν αφορά αυτό την Επιτροπή ανάπτυξη, γιατί το πράσινο κροτήριο είναι μεταξύ εκείνων των χωρών που βρίσκεται στη μεταβατική περίοδο. Δεν είναι δηλαδή ακόμα πλή, πια πλήρως στην ε, συνθήκη ΑΚΕ και όχι ακόμα τελείως αυτόνομες. Ε, βρίσκονται σε ένα διάμεσο στάδιο και γι' αυτό για αυτή την περιοχή ίσως δεν θα ήταν καλό να να αναμειχθεί η Επιτροπή ανάπτυξη, αλλά για άλλε ναι. Ωραία, ωραία. Ίσως εδώ παίζει ρόλο η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αλλά όμω. εάν οργανώσουμε αυτή τη συνεδρία εργασία, θα το κάνουμε για να εξετάσουμε όλες τις συμφωνίε Αλλίας, που επίσης αφορούν την ε, ε Επιτροπή Ανάπτυξης ε, Ο κ. Αλφασίνο, η εισηγητή μας, ήσασταν μεταξύ εκείνων ε, της Επιτροπής Αλίας που πήγανε στην Ισλανδία. Γιατί είχαμε μια αντιπροσωπεία στην Ισλανδία, τις οποίες προέδρευσε ο Γκέραν Φέρν, και υπέφεραν μια ε, γραπτή έκθεση που δέχτηκαν όλα τα μέλη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και που μας παρουσίασε ο κ. Φέρν χθε το απόγευμα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στην παρουσίαση αυτή του κ. είναι ότι η αντιπροσωπή αυτή εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα της πολιτικής αλληλείας της Ισλανδίας ότι οι Ισλανδοί στις διαπραγματεύσεις, στις προκαταρτικές για ενδεχόμενη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητούν καθόλου ενίσχυτη στην ε, Αλία ή να είναι μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αλίας και θεωρούν ότι στα ύδατα που οικονομικά ελέγχουν κατάφεραν να εισαγάγουν μια πολιτική που προστατεύει τις πηγές, δηλαδή οι αλείς τους είναι πλούσιοι και τα, οι χθείς τους είναι ευτυχείς. Ας με ελέγξει ο Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα μεταξύ των φίλων της Ελίας και των φίλων των ηχθείων σε αυτή τη χώρα. Και το λέω αυτό στον κύριο Αλφονσίν, γιατί ίσως άσχετα από συμφωνίες συνεργασίες υπάρχουν κάποια διδάγματα που μπορούν να ε, να προσφερθούν από άλλες χώρες. Προτείνω για την έκθεση αυτή γνωμοδότησης να ορίσουμε για τις 30 Ιουνίου την προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. Θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε εμείς την γνωμοδότηση Συνεδρίας Επιτροπής Προπολογών 12 και 13 Ιουλίου γνωρίζοντας ότι η επισουσίας αρμόδια επιτροπή Ηλίας θα συνεδριάσει 31 Αυγούστου και θα μπορέσει να περάσει στην πρώτη δεύτερη σύνοδο του Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια. Τώρα θα μπορέσουμε να περάσουμε στην παρουσίαση και ψηφοφορία της έκθεσης Μπάρμπαρα Ματέρα για την κοινοτοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση προς όφελος, το σημείο 18 λέω, και 19, προς όφελος λέω δύο επιχειρήσεων στη Δανία και οι δύο. Αφενός το ναυπηγείο στην Οντένσε και από την άλλη μεριά μια επιχείρηση της Glass Fiber Company. Θα έλεγα η Μπάρβαρα Ματέρα, η συζήτριά μας, να μας κάνει την παρουσίαση αυτών των δύο φακέλων πρωτού περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ κύριε Ματέρα. Ε, βρίσκομαι κάπω ξαφνιασμένη διότι έκανα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη φορά την παρουσίαση στην Επιτροπή Προπολογισμών. Σήμερα έπρεπε να επικεντρωθούμε επί ψηφοφορία. Όμως δράτω με τις ευκαιρίες που μου δόθηκε για να μπορέσω να πω ότι παρουσιάστηκαν διάφορες τροπολογίες διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά το ΣΥΠΙΑ, το ναυπηγείο, διότι υπήρξαν δύο αιτήματα κινητοποιήσεως του Ταμείου από τη Δανία, αλλά ήταν έτοιμα βασικά από την πλευρά της ΣΥΠΙΑΡΤ που δημιούργησε κάποιες συζητήσεις. Εγώ σε αυτή την περίπτωση ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό το Ταμείο δεν αναδιαθρώνει επιχειρήσεις, δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι που προστίθεται στις κρατικές βοήθειες, διότι βοηθά την ένταξη την επαγγελματική των εργαζομένων, ε, τους δίνει όλες τις δομές στο υλικό και θα πληρώσει και τους ίδιους τους ε, καθηγητές για αυτά τα μαθήματα που οι εργαζόμενοι ε, θα παρακολουθούν για να μπορέσουν να έχουν καινούργιες επαγγελματικές ε, δεξιότητες. Ένα ταμείο που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι βοηθά προσωπικά τους θεωρείται ad personam και δεν βοηθά την επιχείρηση. Όπω κατά το παρελθόν όμω, επειδή κατά το παρελθόν ετέθησαν διάφορε αμφιβολίε, ε, στι επόμενε εκθεσ... αυτού του ταμείου θα προβλέπεται ένα τμήμα που θα εξηγείται οι λόγοι για τους οποίες η συγκεκριμένη εταιρεία Χ και το κράτος μέλος Ψ ε, ζήτησαν την κινητοποίηση αυτού του ταμείου. Αυτό διότι όλοι μας υποστηρίζουμε την αρχή της αφήνειας, της διαφάνειας, ε, της, του όλου εγχειρήματο. Θα υπάρχει αυτή η προστίκη που θα βρουν οι συνάδελφοι στα επόμενα report όσον αφορά το Ταμείο της ε, Κινητοποίησης. Κατά λοιπά, όπως έλεγα, ήδη έδωσα τις λεπτομέρειες την περασμένη φορά, την περασμένη συνεδρίαση, στην περασμένη συνεδρίαση Επιτροπής Προπολογισμών. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ματέρα, εν τω μεταξύ, από ό,τι μου λένε, ε, λάβαμε και άλλους φακέλους. Είχατε εντύπωση να εξάσετε, όχι, όχι, ωραία για που είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε... Εντάξει, όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να σα ζητήσουμε να σχολιάσετε ένα φάκελο που δεν έχετε πάρει. Λοιπόν, προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία. Να. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, oui. Donc nous sommes. Euh, donc nous sommes. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε γνωρίζοντα ότι ταυτόχρονα η Επιτροπή Απασχόληση ε, ψηφίζει αυτή την ίδια στιγμή. Είναι σε επαφή όμω η συγγετριά μα με την Επιτροπή Απασχόληση. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικέ πολιτικέ διαφορέ και αντί να χάσουμε χρόνο, περιμένοντα τον αντιπρόεδρο τη Συρβία, που μου λένε ότι προσγειώθηκε και βρίσκεται καθοδόν μεταξύ αεροδρομίου και κοινοβουλίου και θα φτάσει σε μερικά λεφτά. Λοιπόν, λέω να πάρουμε την ε, λίστα ψηφοφορία για τι δύο εκθέσεις. Θα αρχίσουμε από την έκθεση για την ναυπηγεία, το Odense Steel Shipyard, τροπολογία 4 του κυρίου Χαρτόγκ. Η συγγετρία είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Τέσσερις κατά. Περισσότερες τέσσερα αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Παλτσίτη. Συγχύτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Μία αποχή. Μία αποχή. Εγκρίνεται. 6. Αυτό. Για διαγραφή τη παραγράφου 2. Συγχύτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Τέσσερις κατά. Αποχές. Attention, l'amendement est rejeté. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Αρτόγκ. Ο μπλοκ την 7 και τη 10. Κατά. Αποχές. Με την ίδια ε, πλειοψηφία. Οι δύο αυτές τροπολογίες απορρίπτονται. Πάντα το κύριο Χάρτοκ. Τροπολογία 8 για διαγραφή της παραγράφου 4. Η συγκέντρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. 4. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Με τι πλειοψηφίες. εννέα Χάρτον. Υπέρ. Τέσσερι. Κατά. Αποχέ. Η ίδια πλειοψηφία για την απόρριψη. Τροπολογία Ένα. Χάρτον. Υπέρ. Τέσσερι. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία δύο χαρτών για μία παράγραφο. Εισηγείται έναν κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Τελευταία τροπολογία του κυρίου Χάρτον. Α, όχι, συγγνώμη, όχι. Πραγματικά. Καταπίπτει, αλλά μπορούμε να το ψηφίσουμε. Δεν πειράζει. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία αυτή, η είναι κατά. Πάντα τέσσερι κατά, η ίδια πλειοψηφία. Απόχε. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για την τροποποιημένη έκθεση. Ποιο είναι υπέρ τη έκθεση. Και εγώ. Κατά. 20, 20 υπέρ με τον κύριο καρικά. Αφηρημένο ήταν. Ναι. Λοιπόν, κατά. Τέσσερις. αποχέ. Καμία αποχή. Λοιπόν, η έκθεση για την... Για τον αφήγιο Τζοντέντσε εγκρίνεται 20 υπέρ, 4 κατά και καμία αποχή. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της έκθεσης για την επιχείρηση Glass Fiber. Μία μόνη τροπολογία. Μαρτσίτη. Συγγήτρια είναι υπέρ τη τροπολογία Ένα Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Μία ψήφο κατά. Αποχέ. Μία αποχή. Εγκρίνεται η τροπολογία. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο τη έκθεση. Υπέρ. Για να μετρήσουμε. 21 υπέρ. Πώς είναι κατά. Κατά. 1, 2, 3. Abstention. Αποχές. Τέσσερις κατά. Αποχές, καμία αποχή. 21 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και καμία αποχή. Ωραία. Πολύ καλά μπορούμε αμέσω να περάσουμε στην ψηφοφορία για τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων που απαιτεί δύο μεταφορές για να, χρηματοποιηθούν, να χρηματοδοτηθούν οι ε, νησίες αυτές. Η Σιδονία είναι πάλι η, η μα. μας. Δε λέει εδώ. Mm 5 και 2 10. Η εισηγήτρια είναι μάλλον υπέρ φαντάζομαι. Μάλιστα πρόεδρε. Εγώ θα έλεγα να ψηφίσουμε υπέρ. Και θα έλεγα να ψηφίσουμε και τις δύο μαζί μάλιστα. Την 5 και τη 10. Ωραία. Και τις δύο μαζί. Ποιος είναι υπέρ αυτών των δύο μεταφορών των δελείων. Σε 5 και 10. Θα πρέπει να μετρήσουμε. Αφήστε χέρια σας ψηλά παρακαλώ. Qui ε, est contre. Κατά. Δύο. απόχέ. Καμία αποχή. Εγκρίνω λοιπόν αυτέ τι δύο μεταφορέ. 24 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Bien. Je vous remercie. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Εξαντλήσαμε την σε διάταξη. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον αντιπρόεδρο τη Σερβία. Θα έλεγα να διακόψουμε 2-3 λεπτά. Αλλά παρακαλώ να παραμείνετε στην αίθουσα. Από ευγένεια προς τον κύριο Τζότζικ που θα έρθει τώρα. Θα έχουμε ανταλλαγή από μία ώρα και μετά θα τελείξει η συνεδρίαση. Διακοπή μερικών λεπτών. Λοιπόν, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε ξανά. Να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Σερβικής Κυβέρνησης. Τον ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας και τον ευχαριστώ επίσης που δέχτηκε να αλλάξουμε λίγο και το ωράριο δεδομένου ότι τελειώσαμε τις ψηφοφορίες μας πιο νωρίς από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ενώπιόν σας αντιπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η Επιτροπή Προϋπολογισμών συνήθως αντιδρά εξαιτία του ρόλου της παραδοσιακά σε οποιαδήποτε καινούργια δαπάνη. Και προσπαθεί να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των περιορισμένων πόρων που έχουμε ε, σε πολιτικές οι οποίες έχουν υψηλή ορατότητα σε σχέση με τους πολίτες μας. Είμαστε πολύ ανοιχτοί όμως τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πολιτική γειτονία, την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και βέβαια πάνω απ' όλα ε, στην πολιτική διεύρυνσης. Έχουμε παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις στη Σερβία και νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλης της Επιτροπής και να σας ε, επενέσω για τις ε, τελευταίες και τη σημαντική προσπάθεια που έχει καταβάλει η Σερβία να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Αυτές οι προσπάθειες θα διευκολύνουν τη συνέχιση των ε, διαπραγματεύσεων, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Να σας θυμίσω ε, τα βασικά στάδια τα οποία έχουν λάβει δηλαδή η χώρα στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων. Η Σερβία υπέβαλε την υποψηφιά της επισήμως το Δεκέμβρη του 2009 σύμπτωση, ίσω συμβολική, τη στιγμή περίπου που, άρχισε να, που τέθη σε λειτουργία η Συνδίκη Η προσωρινή συμφωνία τέθησε ισχύ το, την 1η Φεβρουαρίου του 2010 και από τότε η Σερβία ε, άρχισε να εφαρμόζει την ε, Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η διαδικασία επικύρωσης αυτής της συμφωνίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ένα αριθμό επιτροπών που είναι συναρμόδιε για να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και κάποια στιγμή η Επιτροπή Προπολογισμών θα γνωμοδοτήσει προτείνοντα ε, ε, στο Κοινοβούλιο τα κονδύλια εκείνα τα οποία χρειάζονται για να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει. Η σημερινή λοιπόν συνάντηση είναι σημαντική για μας, ε, είναι επικαιρή. Γνωρίζουμε ότι έχετε τεράστια εμπειρία πολιτική και επαγγελματική που ξεπερνάει τη Σερβία, είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκή εμπειρία. Συνεπώς θα σας ακούσουμε πολύ προσοχή. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω καταρχήν λίγο γαλλικά για να αλλάξω μετά προς τα αγγλικά. Όπως ξέρετε έχω ζήσει αρκετό χρόνο στη Γαλλία. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση. Δεν συνηθίζεται ένας εκπρόσωπος κυβέρνησης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απευθύνεται σε μια επιτροπή όπως η δική σας. Συνήθως μας καλούν στη γιορτή και στις γιορτές Στι ε, στις δηλαδή εκδηλώσει και στις επιτροπές που έχουν σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις. Ε, βρίσκομαι εδώ όμω αφενός ε, για να κάνω ένα απολογισμό. Έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ στις δημοσιονομικές προοπτικές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να ξέρει σε πού χρησιμοποιούνται τα κονδύλια τα οποία μας έχουν δοθεί και ποιο αντίκτυπο έχουν. Και δεύτερον, ε, θα σας κάνω μια μικρή παρουσίαση της οποίας ο τίτλος ακριβώς ε, είναι ε, προτάσεις για, για το μέλλον. Η Επιτροπή σας και η Επιτροπή Σούρε συζητούν πολύ τελευταία για, τη, για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2013. Και θα σας μιλήσω, κατ' εξαίρεση, όχι μόνο εκ μέρους της Σερβίας, αλλά εκ μέρους όλων των Βαλκανικών χωρών, γιατί ε, τον Απρίλιο στο Βελιγράδι υπογράψαμε μια κοινή θέση, μας τη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς να εξελίσσονται οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο μετά το 2013. Ελπίζω να έχετε στα χέρια σας τρία έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο είναι αυτή ακριβώς η παρουσίαση. Το δεύτερο έγγραφο είναι η επιστολή που εστάλει ε, σε αρκετούς επιτρόπους και περιγράφει τις θέσεις μας. Είναι ένα position paper. Και ένα τρίτο έγγραφο ε, με την ε, ομιλία μου, την αυριανή ομιλία μου. σχετίζεται, αναφέρεται και στη συνεργασία μας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και με τις εργασίες μας ε, για την ε, επίσημη απόκτηση της ε, ιδιότητας του υποψήφιου, της υποψήφιας χώρας. Τώρα θα ήθελα να συνεχίσω στα αγγλικά. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη για τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια σε σχέση με, την, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι εξαιτία της κρίσης ή εξαιτία των επιπτώσεων μπορεί να έχει στην μελλοντική διεύρυνση. Θα είμαι ειλικρινής. Εμείς στα Βαλκάνια γνωρίζουμε ότι μετά την ένταξη της Κροατίας, την οποία καλωσορίζουμε όλοι και επιθυμούμε, η οποία θα λάβει χώρα χώρα γύρω στα μέσα του 2013 από ό,τι φαίνεται, ε, για αρκετά χρόνια δεν θα ενταχθεί καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός ενδεχομένως της Ισλανδίας. Και αυτό το γνωρίζει η κοινή γνώμη. Το ξέρουμε εμεί το ξέρει η κοινή γνώμη. Γιατί ε, ισχύει αυτό. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πολλέ ώρε, Αλλά αρκεί να πω ότι ε, το Βελιγράδι και τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια γνωρίζουν, γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα μακρύ δρόμο μπροστά μα, Με πολλά εμπόδια, με, πολλές, ε, με πολλά απαιτητικά κριτήρια, αυστηρά κριτήρια. Ε, έχουμε Έχουμε λοιπόν πολλά κριτήρια αυστηρά μπροστά μας και δεν διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Ε, ο, πριν από χρόνια ε, είχαμε την ιδέα από την προηγούμενη ε, δεκαετία να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί εποχής Τζίντζιτς Ε, θέλαμε να ξεκινήσει ο 21ος ε, αιώνας με ειρήνη και γι' αυτό το λόγο είχαμε θέσει μετά στόχο του 2014 ως ένα ε, αιώνα μετά το 1914. το χτυχάσαμε και αυτή την προθεσμία και εσείς αναγνωρίσατε από την άλλη μεριά στην έκθεσή σας ότι οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει επίσης να διαρκέσουν 7 έτη. Ε, κατά τη διάρκεια αυτών των 7 ετών, τόσο η Σερβία όσο και τα άλλα Δυτικά Βαλκάνια θα είναι λοιπόν μάλλον εκτό ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα πάει η οικονομία σε αυτά τα χρόνια. Τα προβλήματά μα δεν ξεκίνησαν με τον Μιλόσεβιτ. Οι επενδύσει ε, στι υποδομέ από τη δεκαετία του 70 ήταν ανεπαρκεί. Επίση, έχουμε και διμερεί θέματα, ε, διμερεί σχέσει, οι οποίε έχουν δημιουργήσει ενεργειακέ συνδέσει, αλλά όχι μεταξύ όλων των χωρών. Μετά ε, η, η κατάσταση μας δείχνει ότι αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, ε, οι πιέσει θα αυξηθούν στα Δυτικά Βαλκάνια. Και όπως είπε ο Λαβουαζιέ κάποτε, η φύση ε, φοβάται το κενό. Και αν δεν, έχουμε ως στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχουμε κανένα στόχο. Αυτό είναι ο φόβο. Συνεπώ πολιτικά, οικονομικά και ε, δημοσιονομικά ε, είναι σημαντικό να έχουμε αρκετά εργαλεία έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως η Ευρώπη θα είναι το νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα μας. Αν αναφερθήκατε την ε, παράδοση Μλάντιτς. Εγώ υπέγραψα την ε, Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε ήταν ε, πραγματικά δραματική κατάσταση με το κοσυφοπαίδιο. Οι εθνικιστικές δυνάμεις προσπάθησαν στη Σερβία να πάρουν την κυβέρνηση και να οδηγήσουν τη χώρα μας σε προς άλλη κατεύθυνση. Όμως, ο, η Fiat που είπε ότι ε, θα επενδύσει σε μια Ευρωπαϊκή Σερβία. Ε, ο κύριος ε, Φρατίνη, ο οποίος επίσης μας υποστήριξε εκ μέρους της Κομισιόν, με αυτή τη βοήθεια καταφέραμε και νικήσαμε. Χωρί αυτού δεν θα μπορούσαμε να νικήσουμε και χω, αν δεν είχαμε νικήσει ούτε ο Μλάντιτ ούτε ο, ο θα ήταν στην, στην Χάγη. Ε, ούτε θα είχαμε συλλάβει τους λαθρέμπορους, ε, ναρκωτικούς και, ε, ναρκωτικών και άλλους. δεν θα είχε ψηφιστεί το ψήφισμα για τη Σρεμπρένιτσα που ψήφισε το Κοινοβούλιο. Δεν θα είχαμε καταφέρει να συνδιαχειριστούμε με την Κροατία και τις τρεις κοινότητες της Βοσνίας. δεν θα είχαμε καταφέρει να διαχειριστούμε το, την λειτουργία της Βοσνίας. Συνεπώς, αυτό που σας ζητώ είναι να ε, εξασφαλίσουμε ε, ρεαλιστική υποστήριξη. Δεν ε, εθεροβατούμε. Το 2014 δεν θέλουμε τα Δυτικά Βαλκάνια να ξεχαστούν. Γιατί αν ξεχαστούν, θα ήταν σαν να έχουμε ξεχάσει 20 εκατομμύρια κατοίκους. Ε, δεν είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ε, Ευρώπης, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι, διότι είναι μια περιοχή πολύ περίπλοκη. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τώρα την έκθεσή μου με τα βασικά μηνύματα. Πρώτο βασικό μήνυμα. Χρησιμοποιώ Ποιήσαμε την τελευταία δεκαετία ε, πολύ αποτελεσματικά τα κονδύλια που μας έχουν χορηγηθεί. Τα τελευταία δέκα χρόνια ζήσαμε δύο σημαντικές στιγμές. Πρώτον, μετά την νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων, ε, ζήσαμε δύο χρόνια που χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνθρωποι που έριξαν το Μιλόσεβιτ δεν θα είχαν ούτε φάρμακα ούτε ε, ηλεκτρική ενέργεια. Ε, και εμείς συνεχίζουμε να υπενθυμίζουμε στους πολίτες μας το πόσο πολύ μας βοήθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Το δεύτερο μου μήνυμα είναι το εξή. Η διαφορά ανάμεσα στις πρόσφατα ενταγμένες ε, χώρες και στις ε, χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον είναι τεράστια. Δηλαδή οι, οι, χώρες που εντάχθηκαν το 2004 είναι ε, ε, 10 φορές πιο μπροστά από τις χώρες που ανήκουν στην ε, Συμφωνία της Θεσσαλονίκης του 2003. Όση πολιτική βούληση και να έχουμε, αν δεν υποστηριχθούμε, δεν θα μπορέσουμε να συμμορφωθούμε τα κριτήρια. Τρίτον, μετά το 2013 θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η προνταξική βοήθεια λαμβάνει σωστή προτεραιότητα. Να, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και να βασίζεται σε project τα οποία θα είναι προς κοινό όφελος και πιο πάνω απ' όλα να είναι ρεαλιστική η υποστήριξη αυτή. Θα πρέπει να εντοπίσουμε αυτά τα project που θα είναι προς κοινό όφελος και θα μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε και εσείς εδώ και εμείς εκεί ενώπιον της κοινή μας νόμης. Αν δείτε το χάρτη θα διαπιστώσετε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ε, παρόλο που κάθε χώρα λέει πως είναι στρατηγικά τοποθετημένη, η Σερβία στα Δυτικά Βαλκάνια ε, είναι ο πιο σύντομος δρόμος από τη Βιέννη προς την ε, Κωνσταντινούπολη τις, και τις αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής που μετά την Αραβική Άνοιξη θα γίνουν πιο σημαντικές ενδεχομένω. Τελευταίο μου μήνυμα περιέχει δύο πράγματα. Πρώτον, ε, το να αλλάξουμε μόνο αυτά στα οποία συμφωνούμε όλοι δεν είναι αρκετό. Κοιτάξτε την Κροατία. Η Κροατία παίρνει 150 εκατομμύρια περίπου ευρώ το χρόνο. 60 με 70% αυτών των πόρων, όπως και στη Σερβία, ε, είναι αμοιβέ ε, συμβούλων που ε, ζουν εκεί και μας βοηθούν. Μόνο 30 με 40% αυτών των κονδυλίων ε, φτάνουν στους ε, καθημερινούς πολίτες, στους πολίτες μας. Και μόνο για αυτά μπορούμε να πούμε ότι μας, να δείξουμε στους πολίτες μας ότι μας βοηθά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Κροατία σε δύο χρόνια θα παίρνει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 φορές περισσότερο δηλαδή Και αυτό τι δείχνει, ότι ε, έχουμε ελάχιστους πόρους στην αρχή, προενταξιακά, ε, και μετά ξαφνικά αυτό το ποσό, αυτά τα κονδύλια αυξάνονται τόσο πολύ που δεν μπορούν να απορροφηθούν. Αυτό το σύστημα έχει αποδειχθεί λανθασμένο μέχρι τώρα. Οπότε εμείς προτείνουμε ας κάνουμε τις αυξήσεις γραμμικά, σταδιακά, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προετοιμάσουμε πολύ καλύτερα τα θεσμικά μας όργανα, του θεσμούς μας Και γιατί δεν επιλέγετε εσείς οι ίδιοι, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν, τα project τα οποία πιστεύετε θα είναι τα πιο σημαντικά. Ε, ε, ένταξη των Ρωμά, ενεργειακά σχέδια, σχέδια πανευρωπαϊκών μεταφορών και ε, ε τέτοιου είδους σχέδια τα οποία πραγματικά ε, θα είναι προς κοινό συμφέρον. Αυτή η γραμμική αύξηση το, της προενταξιακής βοήθεια είναι σημαντική. Αν αυτό όμως δεν είναι, δεν είναι δυνατό, αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, ε, θα πρέπει να μιλήσω για κάτι πιο ευαίσθητο. Ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να ανοίξουμε ένα ε, κεφάλαιο ε, για την προενταξιακή βοήθεια ε, στον προπολογισμό για τις υποένταξη ε, χώρες. Το δεύτερο σημείο για αυτό το μήνυμα είναι ότι προτείνουμε να μπούμε στο ευρωπαϊκό εξάμεινο αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν επηρεάζει τις μακροοικονομικές πολιτικές ε, των υποένταξη χωρών. Υπάρχει ένας ε, πολύ καλά οργανωμένος πολιτικός διάλογος για δικαιώματα μειονοτήτων, ε, οικοδόμηση θεσμών κλπ. Αλλά η Ευρώπη δεν επηρεάζει το πώς λειτουργεί ένα συνταξιδοτικό ταμείο στις ποένταξεις χώρες, για παράδειγμα. Έχει η Ευρώπη τα γενικόλογα κριτήρια της Κοπενχάγης, αλλά δεν έχει ένα μοχλό για να επηρεάσει μακροοικονομικές πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο, για να αποφύγουμε οι μελλοντικές υποένταξη ε, χώρες ε, να μπουν τα μελλοντικά μέλη να μπουν με δημοσιονομικά που δεν είναι σε καλή κατάσταση ε, θα μπορούσαμε να μπούμε στο ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο κάτι που θα μας έδινε εγγύηση και για τις αγορές με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε πιο ευθυνή χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να αποφύγουμε ε, ε τις, ε, τα υψηλά επιτόκια ε, που για τα δάνεια τα οποία παίρνουμε από τις δικές μας τράπεζες με πολύ ψηλά επιτόκια τα παίρνουμε αυτά 4, 5-7% θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό λοιπόν ε, οπότε από αυτή την πλευρά εμείς κερδίζουμε εσείς τι έχετε να κερδίσετε τώρα θα κερδίζετε το εξή θα είχατε μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάσετε τα πράγματα. Δηλαδή, ε, ένα τέτοιο χρηματοδοτικό μέσο εγγύησης των Δυτικών Βαλκανίων θα σήμαινε ε, το τέλος του οικονομικού λαϊκισμού στη χώρα μας. Δηλαδή οποιοδήποτε πολιτικός λέει, ε, θέλει να κερδίσει την, τις εκλογές λέει θα αυξήσουμε τους μισθούς και τις συντάξει κατά 30%. Ε, ενώπιον αυτών θα θα υπήρχε το επιχείρημα, αν έκανε κάτι τέτοιο, θα είχαν στην πρόσβαση σε αυτό το Ταμείο Δυτικών Βαλκανίων. Ε, δηλαδή, θα... ένας τέτοιος μηχανισμός θα είχε την ε, δυνατότητα να ευθυγραμμιστεί η οικονομική πολιτική των υποένταξη χωρών με την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Σερβία λοιπόν μετά από 7-10 χρόνια μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα όριο συνταξιοδότησης, ηλικία συνταξιοδότησης περίπου ε, την ίδια με αυτή που θα ισχύει και για την χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μετά από αυτά τα μηνύματα θα μπορούσα να σας, δίσω, να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες διαφάνειες. Όσον αφορά, λοιπόν, το παρελθόν, έχετε διάφορες εκθέσεις. Όχι μόνο για τις εκ της Σερβίας, αλλά και των δικών Βαλκανίων. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη μέχρι τώρα. Περάσαμε δραματικές εποχές, όπως σας είπα. Το 2003, παραδείγματι, όταν ο Πρωθυπουργός μας σκοτώθηκε από τον Όχλο, και το μίσος που στάφει εναντίον μας, καταφέραμε σε μερικές εβδομάδες να πάρουμε μικροοικονομική βοήθεια. Αυτό ήταν πολύ καλό για την σταθεροποίηση του δυναρίου. Όταν λέμε ότι θέλουμε ένα, το διάδρομο 10, το ότι καταφέραμε να πάρουμε 43 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή των όσων καταστράφηκαν ε, το 1999 ε, από τις βομβισμούς των ΝΑΤΟ, όπως είναι η γέφυρα στον Όβησαντ, είναι κάτι που βοήθησε ε, να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, όχι μόνο, ήταν καλό όχι μόνο για μας, αλλά και για την Ευρώπη. Η ορατότητα λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω βγαίνει από αυτά τα προγράμματα. Είναι τεράστια προβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφέρω μια πτυχή, το ΙΠΑΡ που δεν αναφέρθηκε πολύ συχνά, διασυνοριακή συνεργασία. Θα πρέπει να έρθετε και να δείτε τον ενθουσιασμό με τον οποίο ο απλός άνθρωπος, οι απλοί άνθρωποι, οι ενώσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι δήμοι συνεργάζονται βάσει αυτών των προγραμμάτων. Δεν είναι μεγάλα, των 20.000 ευρώ, 50.000 ευρώ είναι, 100.000 ευρώ το πολύ. Αλλά καταφέρνουν να μαζέψουν κόσμο από Σερβία, Σερβική Βοσνία, ε, ε, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κροατία. Ε, έχουμε συμβολική είναι η οικοδόμηση του Βούκοβαρ είναι σύμβολο τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι μπορούμε να καταφέρουμε μαζί με την Ευρώπη. Ε, τι είναι το πιο σημαντικό, ότι έγιναν αλλεπάλληλοι έλεγχοι και χτυπάω ξύλο, δεν ξέρω που χτυπήσω το έδρανο ή το κεφάλι μου, ε, αλλά μέχρι τώρα όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε σημαντική υπόθεση διαφθορά που να ξεσπασέ. Δύο συνελήφθησαν εδώ και δύο χρόνια, ένα εργαζόμενο στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ενοικοδόμηση και άλλο ήταν στην αντιπροσωπεία στο Βελιγράδι αλλά γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά και την φήμη που υπάρχει, τα διάφορα θέματα, αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο καταβάλλουμε προσπάθειες και κάνουμε και εσωτερικούς ελέγχους όσον αφορά τα ευρωπαϊκά χρήματα. Οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτά θα σταματήσει άμεσα η ε, αδίποτε καλή βούληση υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρησιμοποιούμε το ΥΠΑΡ 1 και 2. Αυτό σημαίνει δημιουργούμε θεσμούς σε διασυνοριακό επίπεδο. 30% ε, από τα 200 εκατομμύρια το χρόνο χρησιμοποιούνται ε, για κοινωνικονομικά θέματα. Δεν έχουμε αρκετά προγράμματα σήμερα επί των οποίων μπορούμε να βάλουμε ε, ευρωπαϊκή σημεία. Έχουμε ένα σύστημα για την αποκεντριωμένη διαχείριση των ε, χρημάτων και είμαστε στην πρώτη από τις έξι φάσεις όσον αφορά την όλη διαδικασία που ακολουθούμε και έτσι του χρόνου θα μπορέσουμε ε, να πληρούμε και ε, όλες και τις πέντε προδιαγραφές που απαιτούνται από το τη διάθεση του κονδυλίου αυτού. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, για την τρέχουσα δημοσιονομική προοπτική, τρέχουσα δημοσιονομικές προοπτικές, να βάζουμε μαζί τη Γεωργία και τα Θετικά Ταμεία. Ε, Ευρώπη 12, έχουμε 261 για τα Δυτικά Βαλκάνια, 2084 για την ε, Ευρώπη των 12. Υπήρχε μια διαφήμιση American Express, περίφημη, που έλεγε ότι έχει τα προνόμια τη τον είναι μέλο κανεί τη American Express. Βέβαια, τον είναι κανεί μέλο έχει προνόμια, αυτό δεν, έχει, δεν αμφισβητείται. Το πρόβλημα είναι ότι με τέτοια μεγάλη διαφορά δεν θα πρέπει να εκπλήσεται κανεί από ότι λόγω αυτού και άλλων λόγων υπάρχουν τεράστιες πιέσεις στις χώρες να μπουν το ταχύτερο δυνατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω δεν θα πρέπει να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους χρηματικούς, θα πρέπει να έρθουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αξιών, λόγω προγραμμάτων, λόγω της εγγύησης που δίνει για την ειρήνη, λόγω των προπτικών και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά τέτοια, ένα μονομερε, μονόπλευρο οικοδόμημα κάνει σαν ημέρα εισβολή την ημέρα της προσχώρησης, οικονομικής εισβολής και αυτή δεν είναι υγιεινή προσέγγιση. Δεν θα χρονοτριβήσω, διότι ήδη ανέφερα τα περισσότερα, έχουμε εντοπίσει και αδυναμίες στη χώρα μας. Ε, μία από τις βασικές αδυναμίες είναι και εξή ότι καμιά φορά υποτιμούμε τις προσπάθειες που απαιτούνται, ούτω ώστε πραγματικά να εφαρμόσουμε προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Θέλουμε να ξεκινήσουμε διάφορα πράγματα, σπρώχνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθούμε να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να καταλάβουμε τελικά καμιά φορά ότι δεν έχουμε τα χρήματα για την σωστή ε, αγορά, εξαγορά γεών ή για σωστή αξιολόγηση συνεπειών για το περιβάλλον και άλλα τέτοια συναφή. Υπάρχουν κάποια σημαντικά προγράμματα, ένα-δύο σημαντικά προγράμματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας ρωτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το προτείνεται αυτό χρειάζονται πιο αυστηροί όροι που πρέπει να τίθενται πριν γίνονται αποδεκτά τα προγράμματα, διότι τότε θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι ότι θα υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα. Ε, λοιπόν, και, τι κερδίζουν όλοι, είναι υποφελέ για όλου. Η Σερβία, και δεν είμαι γι' αυτό, είναι μια χώρα που πηγαίνει σύνοδο κορυφή τη Κοπενχάγη για το περιβάλλον, χωρίς να ξέρουμε πόσο διοξίδιο του άνθρακος εκπέμπουμε το χρόνο. Αλλά Λόγω αυτού κάναμε τις μελέτες και τώρα γνωρίζουμε. Είμαστε στην αρχή, τώρα στην περιοχή, ξεκινάμε τις προσπάθειες όσον αφορά τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας όπως η ηλεκτρική ενέργεια. Η γεωργία είναι, παρέχει μεγάλες δυνατότητες αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε σωστή προσέγγιση, απασχόληση, ποιότητα. 19,6% είναι η ενέργεια στη χώρα μου. Και το να υπάρχουν και δεξιότητε των ανθρώπων για τον 21ο αιώνα είναι επιτακτική ανάγκη και όχι για το 19ο αιώνα. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία, χάρη στην ευρωπαϊκή υποστήριξη. ...400 εκατομμύρια ευρώ από διάφορε πηγές για επενδύσεις, επιστήμη, τεχνολογία και υποδομέ. Χωρίς τη στατική τη Ευρώπης του 2020, χωρί την συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς δεν θα είχαμε τη γνώση και το θάρρος ε, να κάνουμε αυτά τα βήματα. Και τώρα που τα κατάφερε η Σερβία και άλλες χώρες στην περιοχή το αποτολμούν. Καλή διακυβέρνηση, δεν χρειάζεται να χρονοτριβήσω επ' αυτού. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα αναφέρω ακροθυγώς, διότι θεωρώ ότι δεν εξαρτάται από εμά από τις υποψήφιες χώρες να εκφράσουν άποψη. Όπως γνωρίζετε όμως, 1% του ΑΕΠ θα παραμείνει ο προπολογισμό από ό,τι καταλαβαίνω. Το Κοινοβούλιο έχει διαφορετική άποψη. Αλλά διάβασα επιστολή των πέντε Υπουργών Οικονομικών και διάβασα και βρετανικές επιστολές και άλλες επιστολές από 12 χώρες συνοχής. Δεν είμαστε προσκεκλημένοι συμμετάσχουν στη συζήτηση. Λοιπόν, αν λέμε ότι είναι 1% του ΑΕΠ η πρόταση ποια είναι. Ότι οι χώρες διεύρυνσης, όχι γειτονία, χώρες διεύρυνσης που συμπεριλαμβάνουν τα 20 εκατομμύρια Δυτικά Βαλκάνια, 300.000 Ισλανδία και 73 εκατομμύρια την Τουρκία. Όλες, όλους μαζί. Μέσα σε ένα εργαλείο. Αυτό δεν είναι καλό. Διότι ε, 3-4% έχουμε αύξηση εμείς, 10% ε, η Τουρκία. Ο πληθυσμό μας μειώνεται, η Τουρκία αυτέ στα 100 εκατομμύρια σε μερικά χρόνια. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διατηρήσει το ΙΠΑ σε ένα, ένα ενίο κομμάτι. Και πρέπει να καλυφθούν διαφορετικές πραγματικότητες και αυτό δεν είναι εύκολο. Αν παραμείνει ως έχει από το 1,3% του προπολογισμού να μειωθούν να μειωθεί στο 1% γιατί μπαίνει η Κροατία, τι σημαίνει όλο το θέμα της διεύρυνσης όχι μόνο πολιτικά αναβάλλεται, αλλά για αυτή τη δεκαετία αντιπροσωπεύει μόνο το 0,01% του ΑΕΠ. Και αντίθετα με άλλους τομείς, η υποστήριξη για τις χώρες της διεύρυνσης ε, ε, εφαρμόζεται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 0,01% συντεριάζει σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να καταλαβαίνετε ποια είναι η απάντησή μου σε αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, λοιπόν, ε, ακόμα και ελάχιστε αλλαγέ στο σύστημα ε, θα έχει τεράστιε συνέπειε επιτόπιε. Δεν μιλάμε για δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εφικτό. Αυτές είναι οι πέντε ιδέες. Ε, γραμμική προσέγγιση να αφορά την κατανομή των πόρων. Ε, να υπάρχουν περισσότεροι συντονιστές είπα, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει το βασικό πλαίσιο συναθρίζοντας διάφορους θεσμούς αλλά δεν, έχω, δεν το είχαμε ακούσει, μας παρουσιάστηκε δεν είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε συμβουλευτικό ρόλο το είπα καθυστέρησε δύο χρόνια όταν ξεκίνησε το MFF. Θα πρέπει να γίνουν επιτυχίε να έρχονται έγκαιρα και μετά έχουμε και την, το μέσο για, την, για τις εγγύσεις Δυτικά Βαλκάνια. Και αξίζει μια εικόνα χίλιας λέξεις, όπως λέμε. Εδώ έχουμε κάτι υποθετικό παρουσιάζουμε. Η, το παρόν σύστημα είναι η γαλάζια γραμμή. Περίπου 200-300 εκατομμύρια και μετά στα 2 δισεκατομμύρια Κροατία-Σερβία. Και η κόκκινη γραμμή είναι αυτό που προτείνουμε. Η ολοκλήρωση, το, η έκταση μεταξύ των δύο καμπύλων ε, θα επιστραφεί στο Κοινοβούλιο σε εσά και τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ. Το ποσό σε αυτή την περιοχή. Ίσως 4 ε, δισεκατομμύρια ευρώ που μπορεί να για το διάδρομο 10. Εμείς δεν ζητήσαμε από την Ευρώπη, τα Δυτικά Βαλκάνια, ούτε ένα ευρώ για να περάσουμε την κρίση. Κάποιες χώρες αύξησαν τους φόρους, η Σερβία δεν το έκανε αυτό, μειώσαμε τις δαπάνες, το έλλειμμά μας θα είναι κάτω από 4% φέτος, θα είναι 3% του χρόνου και έχουμε ένα νόμο για, φορο... για οικονομική ευθύνη... και θα πρέπει να ετοιμαστούμε για τι δημογραφικέ αλλαγέ και να ελέγξουμε το έλλειμμα. Χρησιμοποίησαμε 7 ποσοστέ μονάδε του ΑΕΠ και το χρέος μας είναι 3% το ΑΕΠ. Είναι κάτω από τα κριτήρια του, της Κοπενχάγης, αλλά ο νόμος δεν μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε 4,5%. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης κλπ. Ή θα ζητήσουμε περισσότερα. Αυτή η περιοχή λοιπόν ανάμεσα στο ΔΕΛΤΑ, στο τρίγωνο που χρησιμοποιείται μεταξύ κόκκινης και γαλάζιας γραμμής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει η μακροοικονομική ε, ενίσχυση να γίνει πιο επίκαιρη. Όχι μόνο να χορηγείται όταν έχουμε πλημμύρε. Να είναι κάτι υποφελές για όλους. Εμείς θα έχουμε σταθερούς ε, πόρους, θα προστατευόμαστε από τη διεθνή κερδοσκοπία η Ευρώπη ε, επηρεάζει πολύ τις μακροοικονομικές πολιτικές, έχουν αποτελέσματα μακροοικονομικές πολιτικές και μακροοικονομικά οποιαδήποτε χώρα προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ε, βιώσιμη και οικονομικά και συνταξιδοτικά. Ε, όσον αφορά το έλλειμμά μας, για όλη τη δεκαετία θα είναι 2 μέχρι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά το, στη Σερβία. Και είμαστε περίπου το 60% Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω μετά από όλα αυτά. Ελπίζω να μην χρησιμοποίησα πολύ από το χρόνο σας. Ίσως επειδή είχα τη δυνατότητα για πρώτη φορά τη μεγάλη ευκαιρία να σας μιλήσω, να μακρηγόρησα και αν με ξανακαλέσετε υπόσχομαι να είμαι συντομότερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είδατε ότι οι συνάδελφοι σας χειροκρότησαν αυθόρμητα άκουσαν με πολύ προσοχή την εισαγωγή σας. Ε, αρκετοί συναλφοί έχουν ζητήσει το λόγο. Η παρουσία σας ήταν πολύ σαφής, ε, ευνόητη, ε, η οποία βέβαια ε, γεννά πολλά ερωτηματικά. Καταρχήν ο Γκόραν Φέρμ, που είναι συντονιστής ε, δηλαδή εκπροσωπεί το, το, την ομάδα του σοσιαλιστικού, το, τη σοσιαλιστική ομάδα. Συγγνώμη. Είμαι και συντονιστής της, ε, των μελών του Σοσιαλιστικής Ομάδας στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και εισηγητής για θέματα διεύνησης αυτήν εδώ την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και σας συγχαίρω για την ε, πρόοδο που έχει επιδείξει η Σερβία και στην, σε πολιτικό επίπεδο και στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ορισμένες σκέψεις και ορισμένες ερωτήσεις. Ε, συζητούσαμε την ε, διεύρυνση και με παλιότερα με την ε, Κροατία ή με τις χώρες που μπήκαν το 2004-2007 και θυμάμαι ποια ήταν τα προβλήματα τότε. για παράδειγμα, το δικαστικό σύστημα. Η, ε, αναφερθήκατε στη διαφθορά. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις διαφθορά στη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, όμως η διαφθορά είναι κάτι πολύ πιο πλατή, επηρεάζει όλη την ε, κοινωνία και αποτελούσε πάντοτε πρόβλημα και με τις προηγούμενες πανταξή χώρες. Ε, ε, το Κοινοβούλιο το έφυγε ιδιαίτερα. Και στην, πρόοδο, στην έκθεση πρόοδου του 2010 για τη Σερβία είναι ένας από τους τομείς ε, για τους οποίους η Κομισιόν εξέφραζε επικρίσεις. Η Σερβία έλεγε έχει κάνει πολύ λίγη πρόοδο στην ευθυγράμμιση του δικαστικού συστήματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην διαχείριση της οικονομίας. Δεν ξέρω αν έχετε σχόλια γι' αυτό. Άλλο προ, άλλη ε, περιοχή στην οποία πάντοτε είχαμε προβλήματα είναι η επιδοτή τη οικονομία. Με την Κροατία συζητούμε πολύ τις επιδοτήσεις των αυπηγείων, για παράδειγμα, και βέβαια το, την κληρονομιά ενός κεντροσχεδιασμένου συστήματος, οικονομικού συστήματος, ε, ε, που βασιζόταν σε επιδοτήσεις και στην ε, κρατική κυριότητα ε, των, των αγαθών. Τρίτο πρόβλημα που είχαμε πάντοτε είναι η κατανομή του, του πλούτου στη χώρα. Για παράδειγμα, το Βελιγράδι, άμα το συγκρίνουμε με την Ήπεθρο, πάντοτε οι μεγάλες πόλεις αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, αλλά το θέμα είναι η κοινοτική χρηματοδότηση να χρησιμοποιείται και για την ανάπτυξη πέθρου και για περιφερειακή ανάπτυξη, έτσι ώστε να εξισωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Αυτό ήταν πάντοτε πρόβλημα σε όλες τις καταβάσεις της ε, υποένταξη χώρες στο παρελθόν. Τέταρτο σημείο. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, κοινωνικοί φορείς, κοινωνία των πολιτών και μικρά project ε, μια χώρα που θέλει να αναπτυχθεί γρήγορα συνήθως εστιάζεται σε μεγάλα στρατηγική σημασία project που θα αλλάξουν όλη την κοινωνία. Ε, εμείς όμως πιστεύουμε πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Θα πρέπει να υποστηρίξετε και μικρότερες οργανώσεις, ε, οργανώσεις για την ανάπτυξη πέθρου, μικρότερα project για να ε, αποφύγουμε ε, μία μονομερή ανάπτυξη. Ε, το πρόγραμμα IPA είχε πρόβλημα με την πτυχή του για την, την κοινωνία των πολιτών. Δύσκολα έφταναν τα κονδύλια σε μικρές ε, επιχειρήσεις και μικρές οργανώσεις. Έχετε σχόλια για αυτό το ζήτημα. Ε, τέλος, είναι πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες οι ιδέες σας ε, για την προοδευτική αύξηση, για παράδειγμα, της ε, ενίσχυσης της προενταξιακής βοήθειας. Το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια υποένταξη χώρα και σε μια χώρα που έχει γίνει μέλος. Ε, δεν είμαι εντάξει, δεν αμφιβάλλω ότι η Σερβία έχει αποφασιστεί να γίνει μέλος, οπότε τίθεται θέμα το, για το, ε, το ερώτημα είναι πότε. Πλην όμως υπάρχει πάντοτε μια διαφορά ανάμεσα σε μια υποένταξη χώρα και σε ένα μέλος, σε ένα κράτος μέλος. Η διαφορά βέβαια αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη. Συμφωνώ και δημιουργεί προβλήματα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Η, η, διαφορά αυτή είναι πολύ μεγάλη. Je vous Monsieur Bocroche. Ο κ. Μπόκρος. Καλωσορίζω τον αντιπρόεδρο της σερβικής κυβέρνησης. Ναι, ε, πολύ δραστήριος ε, όλη την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να βοηθήσει τις προοπτικές της χώρας του. Ήταν ε, πολύ χρήσιμη η παρουσίασή σας, τίποτα χειρότερο. Ήταν πολύ καλή η παρουσίασή σας να σας κάνω μερικές έτσι, προκλητικές λίγο ερωτήσεις για να προχωρήσουμε την συζήτηση. Η πρότασή σας για την γραμμική αύξηση ε, το, της ε, βοήθειας προς τα Δυτικά Βαλκάνια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρουσα λέω, δεν λέω αν ότι είναι καλή ή κακή, αυτή τη στιγμή δεν την κρίνω. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο ε, ποια είναι η άποψή σας για το πώς η αυξημένη βοήθεια θα οδηγεί σε καλύτερη οικοδόμηση θεσμών. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα, αυτό είναι το θέμα. Εσείς λέτε βέβαια ότι το εμβαδών μεταξύ της κόκκινης και της μπλε γραμμής πριν την ένταξη είναι μικρότερο από αυτό που ε, ε, από το εμβαδό μετά την ένταξη. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προκαταβολή αυτών των ποσών, των κονδυλίων, για τη δημιουργία καλύτερων θεσμών, καλύτερης διακυβέρνησης και για να δώσετε μεγαλύτερη όθηση στην ε, προενταξιακή διαδικασία. Έτσι ώστε η ένταξη να είναι επιτυχημένη και ενδεχομένως νωρίτερα από ό,τι με τα υπόλοιπα σενάρια. Εγώ είμαι υπέρ της ένταξης όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, έτσι κι αλλιώς με ξέρετε. Διάβασα και το έγγραφο πολιτικής σας και στην ε, πρώτη σελίδα Βλέπω το λόγο και στο τέλος βλέπω και την υπογραφή τεσσάρων χωρών. Αλβανία, Μαυροβούνιο, Μακεδονία και Σερβία. Υπάρχουν και άλλες δύο χώρες. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψη σας για την Βοσνία και για το Κωσυφοπαίδιο. Καταλαβαίνω, το θέμα είναι πολιτικά πολύ ευαίσθητο, οπότε δεν περιμένω ότι θα ε, κάνετε κάποια ε, ριζοσπαστική δήλωση αλλά είσαστε συνεχώς στα φώτα της δημοσιότητας ως πολιτικός, οπότε ε, γνωρίζετε πως ε, αν, πρέπει να, αν θέλετε να μιλάτε εξ ονόματος όλων των Δυτικών Βαλκανίων, θα πρέπει να μιλάτε εκ μέρους όλων, συμπεριλαμβάνουμε της Βοσνίας και του Κωσυφοπεδίου. Οπότε θέλω να πείτε την άποψή σας για τις ε, ε προοπτικές με το Κωσυφοπέδιο ιδιαίτερος. Τέλος, Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτές οι προτάσεις περί γραμμικής αύξησης κλπ. Ε, έχουν συζητηθεί με τον Επίτροπο Φίλε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε και την άποψη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί το θέμα τελικά δεν είναι τα χρήματα. Τα ποσά είναι μικρά, έχετε δίκιο. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, ε, οικοδόμησης θεσμών και μέλλοντος της πολιτικής διεύρυνσης. Σας εύχομαι καλή τύχη. Merci, mon cher collègue. Madame Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Τζέλιτς, καταρχήν θα ήθελα εξ του ΕΛΚΑ να σας συγχαρώ και να εκφράσω την πλήρη μας υποστήριξη για τις προσπάθειες σας και ερευνητικά μηνύματα που στέλνει στους Ευρωπαίους εταίρους. Θα αφαιρθώ στην ανάγκη των ε, υποδομών ε, και τις που καταβάλλεται. Εγώ ε, ήμουν στην υπόθεση στην Βουλγαρία όταν η Βουλγαρία πήρε το καθεστώς της υποψηφίου χώρας. Έχω να σας πω ότι η ευρωπαϊκή πίεση για μεταρρυθμίσεις εν μέρη με οικονομική ενίσχυση είχε σημαντικές επιπτώσεις στις προσπάθειες κινητοποίησης της χώρας μου προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε το ποσοστό της ενίσχυσης στη Βουλγαρία με 30%. Μια ε, βοήθεια της τάξης των 400 εκατομμυρίων ανά έτος προενταξιακά. Αυτά τα ποσά δεν ήταν μόνο σημαντικά για να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους μας, αλλά βοήθησαν την ε, κυβέρνησή μας να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα. Όταν αναγνωριστεί η ευρωπαϊκή προοπτική δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει κανένας προς τα πίσω. Οι εμπειρίες από τη βουλγαρική εμπειρία, ε, το βουλγαρικό παράδειγμα είναι ότι θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα με ξεκάθαρες προσπάθειες συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Προγραμματιστικού Προγράμματος συντονισμού της συνολικής πολιτικής χορήγηση οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων και συντονισμό μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών ο, κυβερνητικών ομάδων. Μπορείτε και Τζέλιξ να μας πείτε πώς εσείς και η κυβέρνησή σας αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά, πώς σκοπίζετε να αντιμετωπίσετε ενδεχομένε ελλείψεις, ιδίως στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να δώσει περισσότερα χρήματα για τις προενταξιακές σας προσπάθειες. Ευχαριστώ ο κύριος Γκοντμανής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Τζέλιτς, θα ήθελα να σας υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την οικονομία σας. Βλέπετε κάποια προβλήματα στο μέλλον άμα γίνετε μέλος. Ή ακόμα το 23% των εργαζομένων σε εσά απασχολούνται στον ενεργοτικό τομέα. Και κάπου το 30% του ΕΠ παράγεται από την ε, ε, Γεωργία. Βέβαια ξέρω ότι είσαστε υπαριθμόν ένα στην παραγωγή φράουλας στον κόσμο που λέτε παντού κατεψυγμένες φράουλες. 25% αλλά βέβαια έχετε επίσης χάλιβα. Αλλά είπατε ότι δεν έχετε εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα πρόβλημα. Υπάρχει κάποια δυνατότητα αναδιοργάνωσης ή όχι. Για τα πέταλα μιλάω τώρα. Και το τελευταίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ζητήσατε βοήθεια για να αντιμετωπίσετε την κρίση. Μειώσατε όμως την οικονομία σας, μειώθηκε κατά 3%, αλλάξατε το νόμισμα. Τώρα από 80 δινάρια περνάει η ισοτιμία στο 64, δεν ξέρω στα πόσα. Είναι ρεαλιστική αυτή η λειτουργία του συστήματος γιατί είχατε μικρή πτώση και τώρα αμέσω επανέρχεστε. Τώρα λέτε ανάπτυξη 5%. Και τι γίνεται με την ανεργία που είναι γύρω στο 14%. Αυτές είναι κάποιες απλές ερωτήσεις προς τα πάνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ρώσο Σουριάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία σας. Θαυμάσια ιδέα να έχουμε μια συζήτηση εδώ και τώρα. Θέλω να σας πω κάτι από τη δική μου εμπειρία που η χώρα μου δεν είναι και τόσο παλιό μέλος, η Ουγγαρία δηλαδή. Πρώτον, περίπου πριν από 50 χρόνια η διακυβερνητική διάσκεψη συζητούσε το θέμα της δυνατότητας της διεύρυνσης και αυτό ήταν μια ανεπίσημη απόφαση. Καλή είναι η διεύρυνση, αλλά όχι με περισσότερα χρήματα. Και άμα κάνουμε μια σύγκριση, τι κέρδισαν οι Πορτογάλοι όταν εντάχθηκαν και τι έγινε με τις χώρες που εντάχθηκαν το 2004, οι διαφορές είναι τεράστιες. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν συνεπείς αυτή τη στάση. Διεύθυνση ναι, περισσότερα χρήματα όχι. Τώρα είναι επικίνδυνο τα λέτε γιατί δεν χρειάζεται περισσότερα χρήματα για τη διεύρυνση. Βέβαια έχετε λίγο πολύ δίκιο. Uh, uh, Ένα πρόβλημα είναι αυτή η γραμμική ανάπτυξη. Αυτό είναι δυνατόν μόνο νομίζω όταν είναι γνωστή η ημερομηνία της ένταξης. Αν είναι άγνωστη η ημερομηνία αυτή, είναι δύσκολο να ζωγραφείς κανένα την καμπύλη σωστά. Αυτό που είπε ο προθεσμός μου τελευταία, νομίζω ότι από ό,τι άκουσα, εξέφρασε τη εμπειρία που είχε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχει κάποια, κάποιος κορευσμός, αν θέλετε, της διεύρυνσης. Πολλά έκανε η χώρα σας βέβαια τελευταία. Πριν από έξι μήνες συζητάγαμε η σωστή με την Ισλανδία, αν ήθελε, και η Κροατία. Και τελείωσε. Και μετά μεγάλη διακοπή. Τώρα αυτά άλλαξαν όλα για διάφορους λόγους και λίγο και χάνει στην Ουγγρική Προεδρία. Γιατί είναι ανοιχτό μυστικό ότι εμείς θέλουμε οι γειτονές μας να βγουν στην Ένωση. Το ίδιο ήταν στο παρελθόν με τη Γερμανία και άλλες χώρες που βρισκόντουσαν στα σύνορα, παρά τα ευχάριστο να καλέσει κανένας τους γείτονες. Εκείθεν. Αν μια χώρα τώρα επιμένει για την ένταξη, βλέπουμε ότι αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός μεταξύ των πολιτών. Από την άλλη μεριά, αν βιαστεί με την ένταξη, πάλι επικίνδυνο είναι. Είναι η οικονομία ανταγωνιστικές επαρκώς για να επιζήσουν στην κοινή αγορά. Αλλιώς θα χάσουμε παραγωγή, θα χάσουμε θέσεις απασχόλησης. Ο εμπορικός ισολογισμός στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ δύσκολος αν δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική η οικονομία μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά χρήματα που υπάρχουν για να μπορέσει να γίνει η οικονομία καταναλωτών ανταγωνιστική, πράγμα που θα επιταχύνει την ένταξή σας που σας εύχομαι να πραγματοποιεί το πληγόρο των δυνατών. Ευχαριστώ κύριο Σαλφόντσι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξετίμησα τα μάλα τα όσα παρουσιάστηκαν που δείχνουν ότι η Σερβία θέλει να προχωρήσει. Και η ομάδα μου και εγώ θεωρούμε ότι τα Βαλκάνια ήδη είναι εντός των συνόρων της Ευρώπης. Είναι περισσότερο λογική ολοκλήρωσης από τη διεύρυνση όσον αφορά τα Βαλκάνια. Θέλουμε να φροντίσουμε ούτω ώστε οι Ευρωπαίοι που είναι στο επίκεντρο του χώρου μας να μπορούν μέσω συγκλήσεως οικονομικής και όχι μόνον Θέλουμε και δημοκρατική σύγκληση και οικολογική σύγκληση και μπορούν να μπουν πλήρω αν τα κάνουν αυτά. Είχατε αναφερθεί στην έλλειψη ανησυχιών ε, όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακος, το κουβέζι του άνθρακος όταν συμμετείχατε στην ε, Σύνοδο της Κοπενχάγης. Βλέπετε τη μεταρρύθμιση θέλουμε. Αν πάρουμε λοιπόν τη φιλοσοφία ότι πρόκειται περί περισσότερο παρά περί εντάξεως, Εν τη αυτή περιπτώση μπορούμε να δούμε την πρότασή σας με ενδιαφέρον για πιο γραμμική προσέγγιση όσον αφορά την διοργάνωση της υποστηρίξεως από πλευράς Ευρώπης προς την πολιτική της ολοκλήρωσης και να φροντίσουμε να έχουμε πιο συνεχόμενα αποτελέσματα, συνεχή αποτελέσματα. Όταν δεν ξέρει κανεί την ημερομηνία προσχώρηση, δύσκολο να προβλεφτεί και να κάνει σωστή γραμμική προσέγγιση. Όσο μιλάμε μια ολοκλήρωση, υπάρχει βεβαιότητα ένταξη. Διότι ε, συνεχίζεται η πολιτική κατάσταση στην, ε, στα Δυτικά Βαλκάνια και αν συνεχιστεί και η βούληση και των κυβερνήσεων των χωρών αυτών να κινούνται προς την κατεύθυνση που περιγράψατε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Και εγώ το βρήκα αυτό πολύ ενδιαφέροντα. Και εμένα αυτό που άρεσε ήταν ότι ήσασταν πάρα πολύ ειλικρινείς γιατί και η δική μου, στη χώρα μου, οι συμπολίτε μα είναι όπω και οι δικοί σα ενδιαφέρονται για τα χρήματα. Και για τα χρήματα μάθαμε σήμερα ότι τα νέα κράτη-μέλη τη Ένωση παίρνουν το δεκαπλάσιο από ότι τα, οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Ανακεφαλή. είπα ότι και οι Γερμανοί το ίδιο λένε. Που όλο λένε, ε, εμείς όλα πρέπει να τα πληρώνουμε. Ακριβώς. η δικοί μου οι, εκλογές δεν θέλουν πια να πληρώνουν. Λοιπόν, αν δεν πληρώνουν αυτοί, ποιος θα πληρώσει. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να ανοιχνεύσετε και άλλες δυνατότητες της οικονομικής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσο εσείς για την ε, ε, περιφερειακή συνεργασία. Πιστεύω ότι πολλά μπορείτε να κάνετε ακόμα. Γιατί δεν υπάρχει μια οικονομική ένωση, γιατί όλα τα κράτη-μέλη έχουν δικό τους νόμισμα, έχουν ε, την ανάγκη θεωρήσεων των διαβατηρίων για πάνε από μια χώρα στην άλλη. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία όπως εκείνη που υπήρξε η Ιουγκοσλαβία πριν από 20-25 χρόνια. Εγώ θα ήθελα οι χώρες των Βαλκανίων να αποδείξουν ότι πραγματικά προτίθενται να συνεργαστούν μεταξύ τους έντονα. Γιατί όταν τα επόμενα χρόνια όλοι στην Ευρώπη ασχολούνται μόνο με το χρήμα, έχουμε χάσει. Δεύτερον, εγώ δεν κατάλαβα Γιατί χρειάστηκατε τόσο χρόνο για να συλλάβετε κάποιους εγκληματίες πολέμου. Και μάλιστα ακούσαμε ότι ορισμένοι από του εγκληματίες πήραν τεράστιες ε, αποζημιώσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να λυθούν αυτά τα προβλήματα και να ε, μπορείτε τίμια να διαπραγματευτείτε μαζί μας. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κι εγώ ένα-δυο δικά μου σχόλια. Στην εισαγωγή σας μιλήσατε γι' αυτό και το ανέφεραν και κάποιοι από τους ομιλητές μετά. Εδώ και κάποιο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί μια κάποιο κόποση ε, διεύρυνσης, κόποση έναντι των διευρύνσεων. Γιατί όταν μιλάμε για συνθήκες διεύρυνσης ε, είναι σαν να μιλάμε <laughs> για μια διεθνή συνθήκη η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από 27 κοινοβούλια πριν αρχίσει να ισχύει. Θα δούμε την Κροατία, και ενδεχομένω και με την Ισλανδία πώ είναι η κατάσταση στην κοινή γνώμη στα 27 κράτη-μέλη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να πείσουν όχι μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και τις 27 κυβερνήσεις και τα 27 εθνικά κοινοβούλια. Το είπατε κι εσείς ε, από την αρχή ότι ε, η διαδικασία αυτή θα αργήσει να ολοκληρωθεί. Η άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι η εξή. Η καμπύλη σα, την οποία ονομάσατε ε, σταδιακή αύξηση, γραμμική αύξηση, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βέβαια, όπως είπε και κάποιος από τους θα ήταν πιο εύκολο να τη δούμε, να την οπτικοποιήσουμε, αν ξέραμε ποια είναι η ημερομηνία ένταξης. Αλλά Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Όλες οι χώρες οι οποίες, οι συνάδελφοι από χώρες οι οποίες εντάχθηκαν πρόσφατα ε, είδαν εξής, το εξής πρόβλημα, αντιμετώπισαν το εξής πρόβλημα. Ε, υπάρχει μια ε, έλλειψη αντιστοιχίας ανάμεσα στην περίοδο που η ενίσχυση είναι μικρή σχετικά, αλλά που, προσθέτω, είναι σημαντική η παρουσία της ε, Διοικητική βοήθεια μέσω προσωπικού τη Κομισιόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο και μετά στο Βελιγράδι και διαφορά λέω ανάμεσα αυτή την περίοδο και ξαφνικά στην επόμενη περίοδο που υπάρχει μεγάλο, υπάρχουν μεγάλα κονδύλια διαθέσιμα για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστρέφει με το προσωπικό της στις Βρυξέλλες και αφήνει μια ντουζίνα ανθρώπων με πολύ διαφορετικό ρόλο πια. Υπάρχει μια αντιστοιχία, μια έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα σε αυτές τις δύο ε, περιόδους και τα πρώτα χρόνια μετά την ένταξη είναι πολλές φορές δύσκολα. Γιατί υπάρχουν πολλοί πόροι, αλλά υπάρχουν και πολλά προγράμματα, τα πρέπει να ελοπιθούν, πολύ, ένα μεγάλος όγκος νομοθεσίας πρέπει να ε, ενταχθεί στην εθνική νομοθεσία, χωρίς να υπάρχει αρκετό προσωπικό και αρκετή εμπειρογνωμοσύνη. Σε χώρες οι οποίες διαθέτουν μια, ένα διοικητικό μηχανισμό ε, ε, με επαρκή προσόντα και τίμιο ε, είναι πιο εύκολο. Σε άλλες χώρες είναι πιο δύσκολο. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πρώτα σε αυτούς τις πρώτες ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά το δικαστικό σύστημα. Όταν ε, πριν από τρία χρόνια συζητήσαμε την κυβέρνηση, ένα από τα βασικά σημεία τα οποία συζητήσαμε στη συμμαχία μας, στον κυβερνητικό συνασπισμό, είναι ότι ταυτοχρόνως θα πρέπει να πολεμούμε και το οργανωμένο έγκλημα και να βελτιώσουμε το δικαστικό σύστημα. Το καθένα αυτά από μόνο του δεν ήταν αρκετό, γιατί είχαμε την ε, εμπειρία των 10 προηγούμενων ετών που είχαμε συλλάβει σοβαρούς εγκληματίες, αλλά το δικαστικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο. Οπότε ασφαλώς το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αφιέρωσαμε μεγάλους, μεγάλα κονδύλια ε, στην ε, καταπολέμηση των λαθρεμπορίων ναρκωτικών και στην αναζήτηση το, του Μλάντιτς και του Χάτζιτς. Ευτυχώς ο Μλάντιτς είναι στο ε, ποινικό δικαστήριο, μας λείπει ο Χάτζιτς μόνο. Ε, έχουμε ειδικέ μονάδες στην αστυνομία μας ε, και ε, ε, ειδικά τμήματα στα δικαστήριά μας που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που να ειδικεύονται στα μεγάλα ψάρια. Γιατί αν δεν συλλάβουμε αυτούς δεν μας πιστεύουν κιόλα και δεν μιλώ για σας. <laughs> Μιλώ για τους πολίτες της Σερβίας. Ο, μας ρωτούν τη χώρα την κυβερνούν αυτούς που αυτοί που ψηφίσαμε ή οι μεγιστάνες του πλούτου και οι ε, εγκληματίες. Αυτό είναι η ερώτηση που μας θέτουν. Και στόχος μας είναι, και αυτή είναι και η, η, δέσμευση του Πρόεδρου μας ε, και, και η υπόσχεσή του, είναι να ε, προχωρήσουμε, να προδέχουμε και σε αυτό. Ο επικεφαλής της ε, Αμερικανικής DIA ήρθε στο Βελιγράδι πριν από ένα χρόνο ακριβώς για να επενέσει ε, τις προσπάθειές μας. Γιατί μέσω της διεθνούς συνεργασίας καταφέραμε και συλλάβαμε, ε, κατασχέσαμε 5 τόνους κοκαίνης στην Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Και ε, δεδομένου ότι έπεσαν τα μεγάλα κεφάλια, άρχισαν και τα πλοκάμια της ε, οργάνωσης να πέφτουν και την περασμένη εβδομάδα στη Βραζιλία ε, κατασχέσαμε καινούριε προσπά... Ε, ε, και στην Ιταλία, τη Γερμανία και την ε, Γαλλία στη Δυτική Ευρώπη. Οπότε αυτό δίνει μια όθηση γιατί με αυτόν τον τρόπο και οι αστυνομίε των άλλων χωρών μοιράζονται πιο εύκολα πληροφορίες με τις δικές μας αστυνομικές αρχές, ε, αυξάνεται η εμπιστοσύνη και στις αστυνομικές αρχές και στο δικαστικό μας σύστημα. Γιατί δείχνουμε ότι υπάρχει πολιτική κάλυψη. Για το δικαστικό λοιπόν σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι περίπλοκο, γιατί στη δημοκρατία υπάρχει ένα ένας χωρισμός ο ε, διαχωρισμός των εξουσιών. Εγώ είμαι ο μόνος της κυβέρνησης Τζίντζιτς που είμαι ακόμα στην κυβέρνηση. Ξανά στην κυβέρνηση μάλλον. Και θυμάμαι από παλιά μιλούσα με τους επικεφαλείς της δικαιοσύνης και τους έλεγα παρακαλώ πολύ βάλτε τάξη στα του οίκου σας. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για σας να διώξετε τα σάπια μήλα αυτούς που έχουν διοριστεί με πολιτικά μέσα, ε, ε, ή τους διεφθαρμένους. Δυστυχώς δεν συνέβη. Σας ομολογώ ότι δεν συνέβη αυτό. Και ο Τζίντζης δολοφονήθηκε εν, εν μέρη. Τέλος θα μας πάρει πολλή ώρα. Αν σας, για να σας το εξηγήσω, ίσως με μια μπυρίτσα ή ένα ποτήρι κρασί. Ε, αλλά δύο από την ομάδα που τον σκότωσαν αφέθηκαν, ε, είχαν αφαιθεί ελεύθεροι από τους εγγελείς παρόλο που είχαν συλληφθεί δύο εβδομάδες πριν. Οπότε θα πρέπει ε, να προσέξουμε πάρα πολύ το δικαστικό μας. Ε, και ξέρω ότι οι Ευρωπαίοι μας βλέπουν ε, υπό το πρίσμα του εγκλήματος. Δεν θέλουμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Είναι ε, ένας λεκές. Όπως λεκές ήταν και ο Μλάντιτς. Ε, γι' αυτό το λόγο κοιτάμε τις χώρες που έχουν ενταχθεί τελευταία και πράγματι είχαν όλες πρόβλημα με αυτό το ζήτημα. Και λέμε, εμείς θα προσπαθήσουμε πιο πολύ για αυτό το ζήτημα και για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που έτσι και αλλιώς πρέπει να πηγαίνουν νωρίτερα και για να ε, γλιτώσουμε από αυτό το λεκέ, ε, από αυτήν την αμάυρωση της φήμης μας. Ε, και βέβαια και για τους πολίτες μας είναι καλό διότι θα πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να στηριχθούν σε μια καλή λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Θα σας στείλω μια παρουσίαση για το πού βρισκόμαστε στη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο νέο σύνταγμα ε, ένα από τα ευαίσθητα σημεία ήταν ο διορισμός των δικαστών και των εισαγγελέων. Ε, όλοι αυτοί ε, διορίστηκαν και χωρίς να μπω στην, σε λεπτομέρειες είναι ε, ότι προσπαθούμε να κάνουμε το λιγότερο, το μικρότερο δυνατό αριθμό λαθών στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο το, η αντιπροσωπεία της εκτελεστικής εξουσίας είναι πολύ μικρή, το ίδιο και στο εισαγγελικό γραφείο, στην Γενική Εισαγγελία, ε, αλλά ε, ε, ήδη η μισή μας προσπάθεια είχε αφιερωθεί σε αυτό. Τώρα στη διαφθορά. Έχουμε ε, την 35χρονη ε, την 35 υπουργό δικαιοσύνης ε, που παρόλο που γέννησε τελευταία δύο παιδιά κυνηγάει τη μαφία, ο από 5-6 σωματοφύλακες συνεχώς, έχει διοριστεί συντονίστρια η καημένη της καταπολέμησης της διαφθοράς Έχουμε ένα ειδικό ε, σώμα και το γνωρίζω πολύ καλά ότι η διαφθορά μειώνεται στη Σερβία. Ε, συλλάβαμε πέντε πανεπιστημιακούς καθηγητές γιατί ζητούσαν δωροδοκία από τους φοιτητές τους και τους έχουμε σε βίντεο. Ε, συλλάβαμε τον επικεφαλής του Ογκολογικού Ινστιτούτου Βελιγραδίου ε, με, να ζητάει δωροδοκία από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Ε, ένας ε, δήμαρχος μεγάλης ε, πόλης συνελήφθη γιατί πουλούσε φτηνά γη η οποία αμέσως μετά ε, έμπαινε στο σχέδιο πόλης και μπορούσε να οικοδομηθεί οπότε αυξανόταν πολύ η αξία της. Ε, ε, όλα αυτά τα κάναμε και σιγά σιγά προχωράμε. Έχουμε κάνει σημαντική προ, πρόοδο και στη μικρή και στη μεγάλη διαφθορά. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το ζήτημα τα επόμενα χρόνια γιατί δεν είναι εύκολο να πετύχουμε. τώρα προσπαθούμε να προλάβουμε και όλες τις καταστάσεις. και με την ε, Transparency International και με την, τον φορέα που έχουμε εμείς για την κατάμυνση διαφθοράς προσπαθούμε να διαπιστώσουμε πού είναι οι αδυναμίες του συστήματος. Ε, έτσι ώστε να μην δίνουμε τη δυνατότητα στους ε, κρατικούς λειτουργούς να διαφθέρονται. Η Σερβία είναι, η Σερβία είναι από τις λίγες χώρες που όλες οι αποφάσεις εμπορικών δικαστηρίων ανεβαίνουν στο ίντερνετ. Ε, με το σκεπτικό τους. Ε, αυτά για τα δύο πρώτα ζητήματα, δεν θα πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ε, η καταπλέμψη του εγκλήματος και της διαφθοράς είναι πολύ σημαντικό, σημαντική και η συνεργασία. Για τις επιδοτήσεις, κάτι που ξέρει ο κ. Μπόκρος, γιατί ήταν συμβουλός μας πάνω σε αυτό, λοιπόν ήταν, είμαστε μία από τις χώρες που αποφάσισε να μην δώσει επιδοτήσεις στο τραπεζικό σύστημα κλείσαμε 80% των στοιχείων ενεργητικών των τραπεζών το 2002 και παύλα, διότι η εμπειρία έχει καταδείξει ότι επανακεφαλοποίηση των α, τραπεζών δεν έχει νόημα. Και απόδειξη είναι ότι 90% στοιχείων ενεργητικού ε, κατέχουν τράπεζες που εδρεύουν στην Ευρώπη και έχουν καλύτερα κεφάλαια από ό,τι στι ε, έδρε του, διότι είναι τέτοιος, τέτοια νομοθεσία. Δεν χρειαστήκαμε το ευρώ για να επανακεφαλοποιήσουμε μετά την κρίση. Όσον αφορά τι επιδοτήσει λοιπόν και τι ενισχύσει, η Σερβία επί 10 χρόνια ακολουθούσε φιλοσοφία να μην ε, προσπαθεί να ζωγονήσει κάτι που δεν μπορεί να ζήσει. Ίσως θα μπορούσε να σε επικρίνεται διότι παίζουμε το παιχνίδι προσέλκυση των επενδυτών και δεν είμαστε οι μόνοι για να προσελκύσουμε την Fiat να φτιάξει ένα εργοστάσιο ενός δις που θα παράγει 250.000 αυτοκίνητα που είναι η απάντηση στην Τάτσια από ό,τι καταλαβαίνω και ένα μοντέλο για την αγορά Chrysler την Αμερικανική έπρεπε να επενδύσουμε 300 εκατομμύρια ευρώ δεν τα δώσαμε στη Fiat τα επενδύσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Είναι μεγάλη ανταγωνισμό διεθνή για τέτοιου είδου προγράμματα και παρέχουμε επιδοτήσει, ενισχύσει και ωφελήματα για, στον κόσμο για να ανοίξουν εταιρείε στη Σερβία. Επιχειρήσει. Όσον αφορά τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, ε, εκείνοι που έρχονται στη Σερβία εκπλήσονται πολύ για το, μεγάλο, για το υψηλό επίπεδο εκείνων που δουλεύουν στι μη κυβερνητικέ οργανώσει στη Σερβία είναι παραπροϊόν της εποχής Μιλόσεβιτς. Πολύ καλά εκπαιδευμένοι άνθρωποι με πολλές δεξιότητες και ακαιρεότητα αποφάσισαν να μην επιρετούν αυτό το καθεστώς και πολύ συχνά επειδή μερικοί από αυτούς ήταν καθηγητές και εκδιώχθηκαν από τα πανεπιστήμια, πολλοί από αυτούς έγιναν ηγέτες με κυβερνητικών οργανώσεων και παρέμειναν εκεί. Οπότε είναι πολύ ζωντανή η σκηνή σε αυτό το τομέα και αυτό που είπατε ναι, κανόνες περί χρηματοδοτήσεως ή κανόνες για χρηματοδότηση μη κυβερνητικής οργανώσεως από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περίπλοκη. Από την ΕΠΑ παίρνουμε 2 με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον τομέα των κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, πέρσι τον Νοέμβριο, για να τι βοηθήσουμε, δημιουργήσαμε ένα γραφείο για σχέση με κυβερνητικέ οργανώσει που εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό και υποψήφιο που επελέγει είναι μια γυναίκα από τον τομέα των κυβερνητικών οργανώσεων και αναπτύσσουμε το σύστημα για να βοηθήσουμε. Θέλουμε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να μπορούν να παίρνουν πόρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αλλού. Επίση, Έχουμε γραφείο για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που έχει συνάψει συμφωνίε σχεδόν με όλου τι μεγάλε μη κυβερνητικέ οργανώσει στη χώρα και νομίζω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι ένα συγκριτικό όφελο για τη Σερβία. Αν κάποιο δημόσιο υπάλληλο δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ε, ε, Τέλο πάντων, μπορώ να σα παρουσιάσω διάφορε μεταρρυθμίσει που κάναμε στου διάφορου τομεί, διότι είχαμε το σύστημα των μη κυβερνητικών οργανώσεων πάντα, που πίεζαν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει στο σύστημα ευθυγράμμιση τώρα, ευθυγραμμισμένη προσέγγιση. Πρέπει να δώσω πολλές απαντήσεις. Μακάρι να ήξερα ποια χρονιά θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γνωρίζω. Και ο κανόνας του παιχνιδιού ποιος είναι, ότι κανείς δεν θέλει να πει πότε. Κανείς δεν γνωρίζει. Άρα δεν θέλουμε να δούμε τα ΜΕΘΕΘ 2014-2020 και να ξέρουμε ότι το πολιτές πλαίσιο έχουμε Σερβία 2018, άντε Μαυροβούνιο 2017 να κάνουμε τέτοιες μαντεψίες. Όχι, ποια είναι η βασική ιδέα. Πιο περίπλοκη, πιο ανεπτυγμένη. Λέμε, ας μην περιμένουμε μέχρι να μπούμε για να αλλάξουμε αυτά που πρέπει να αλλάξουμε. Ε, αλλάζει όλος ο κόσμος, μέρα, νύχτα. Άσχημα πριν, όχι τόσο καλό όσο περιμέναμε μετά. Θέλουμε μια σταδιακή προσέγγιση, όχι μια νυχτή. Σαν έναν έφηβο που μεγαλώνει άλλη υποστήριξη θέλει στα 13, 15, 18. Και, και ακόμα και όταν είναι 20 χρειάζεται υποστήριξη. Τα ξέρω εγώ καλά αυτά. Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη υποδιέρεση μεταξύ υπείων και λιγότερο υπείων προγραμμάτων και μέτρων. Τα πιο επιτυχή προγράμματα δεν είναι αυτά που δίνουν 12 εκατομμύρια ευρώ κατακαιρματισμένα για δημιουργία δυναμικού. Αυτά δεν λειτουργούν εάν δεν συνδέονται με προσμετρήσιμη συνέπεια για τη ζωή των πολιτών. Δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν τα πάντα. Στο δικαστικό τομέα μπορεί να δώσει κανεί στατιστικά στοιχεία. Αριθμό αποφάσεων από τα πρωτοδικεία, περιπίν, που ανετράπησαν. Πόσα δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσει, ποιε εκκρεμούν, με ποια ταχύτητα διεκπεραιώνονται υποθέσει. Ε, τι καθυστέρηση σημειωθεί, πώ έχουν συσσωρευτεί και περιμένουν να εκδικαστούν. Ε, τι γίνεται με τις, ε, ποια είναι η αξιολόγηση εκείνων που χρησιμοποιούν το δικαστικό μας σύστημα. Μπορεί να κάνεις κάνει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ποιο είναι ο σωστός τρόπος. Πολυετή προγράμματα, ήπια και σκληρότερα, που μπορούν να μαδοποιηθούν και μπορώ να δώσω παραδείγματα. Δικαστικός τομέας, οδικό σύστημα δεν θα πρέπει να δείτε συγχρηματοδότηση να κατασκευάζονται δρόμοι. Έχουν και αυτοί που το λένε, αν ο μεταρρυφορικό μα τομέα ε, μολύνει ή δεν προσαρμόζεται όπω πρέπει στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Απ' την άλλη, κίνητρα για την αλλαγή στον ενεργειακό τομέα, να αλλάξουμε το ήπιο τμήμα, είναι περισσότερα τα κίνητρα αν δεν έχουμε. Ε, είναι πιο δύσκολο να προχωρήσουμε στο ήπιο κομμάτι αν το σκληρό δεν προχωρά. Για τη σταδιακή προσέγγιση. Για... Τι λέει η πρότασή μα. Λόγω της κόπωσης που ανέφεραν οι ευρωβουλευτές και ο πρόεδρος, ξέρουμε ότι υπάρχει κόπωσης. Είναι χειρότερη εποχή να ετοιμάσει κανείς πολιτές πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Αλλά για μας τι είναι σημαντικό, να μπορέσουμε να έχουμε γραμμική αύξηση. Όχι με μηχανικό τρόπο. Δεν πρέπει να γίνει μηχανικό τρόπο. Δεν πρέπει να είναι 20% κάθε χρόνο εξάρτητα το συμβαίνει, 20% ή κάτι άλλο. Πρέπει να συνδέεται με την πρόοδο. Κεφάλαια που άνοιξαν αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλου να πούν «Α, μα αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μεγαλύτερη δυναμική». Χρειάζονται ενδιάμεσα κατόφλια, ούτω ώστε η όλη διαδικασία να γίνει πιο ζωντανή, να έχουμε περισσότερα εμπόδια να ξεπεράσουμε, παρά να έχουμε κάτι ανοιχτό για μια δεκαετία πιθανότατα δεν θα προσχωρήσουμε. Αν δεν αλλάξει τίποτα στο κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά με την Ευρώπη, θα πρέπει να τα καταφέρουμε μόνοι μα. Έτσι βλέπουμε τα πράγματα. Και βέβαια θέλουμε να συζητήσουμε περισσότερο λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτή την προσέγγιση. Τώρα για την ολοκλήρωση, για την ένταξη, συμπερίληψη. Οι, Βόσνοι, Βόσνοι φίλοι μας ήρθαν στη συνεδρίαση και είπαν σας υποστηρίζουμε, στείλαν και επιστολή υποστήριξη. Αλλά επειδή δεν έχουν κυβέρνηση ακόμα, ελπίζω σύντομα να αποκτήσουν, δεν μπόρεσαν να έχουν κάποιον εξουσιοδοτημένο υπογράψει. Συμφωνούν όμως. Όσον αφορά το 25ο, στη Ουάσιγκτον, στα περιθώρια τη συνεδρία τη Παγκόσμια Τράπεζα του Ισού Ταμείου, είδα τον νέο συνάδελφο του Κωσυφοδίου επιφορτισμένο για οικονομία και οικονομικά, συζητήσαμε και θα είδατε το έγγραφο. Το έγγραφο είναι ανοιχτό προ έγκριση από άλλου δικαιούχου επίση. Άρα είναι με το παραπάνω πρόσδεκτη να το εγκρίνουν. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε στη Σερβία. Ξέρετε, δεν αναγνωρίζουμε το Κωσυφοπαίδιο ούτε πέντε κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να υπογράψουμε ένα έγγραφο ε, μια οντότητα που δεν αναγνωρίζουμε. Βέβαια, μπορούμε να υπογράψουμε από την Ούνμη κοσυφό Αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι. Η Σερβία επέβαλε ένα ψήφισμα στο, στο, στο ΟΗΕ και ζήτησε να γίνει διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνας. Έγιναν τέσσερι γύροι διαλόγου τον Ιούνιο υπό την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ε, κυρίω υπό την αιγίδα του κ. Κούπερα, την ομάδα τη κυρία Άστον, ελπίζουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Σα αναφέρομαι στην τυφέ σα, δώσω λεπτομέρειε, θα σταματήσω εδώ όμω. Και σίγουρα δύο πράγματα θέλουμε να καταφέρουμε φέτο να λύσουμε. Πρώτα, τα τελωνιακέ φραγίδε, έχουμε πρόβλημα με την ΕΖΕΣ και μετά εκπροσώπηση του Κωσυφοβεδίου σε περιφερειακό αμορφώματα, γιατί σήμερα δημιουργεί προβλήματα και για εκείνου και για εμά και για όλου η Σερβία ε, δεν αναγνωρίζει τη μονομερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας, θέλει να επιληθεί το πρόβλημα, δεν θέλει μια παγωμένη σύραξη, σύγκρουση, ξέρει ότι δεν μπορεί να μπει η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν επιληθεί το πρόβλημα, δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόβλημα με σύνορα και κυριαρχία. time, Ταυτόχρονα ε, είναι και το θέμα της ε, Πρίστινα Λοιπόν, έχουμε κίνητρο. Θέλουμε να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε ιστορικού συμβιβασμού μεταξύ Σέρβων και Αλβανών στο Πεδίο, Διότι τα προβλήματα δεν ξεκίνησαν και με τον Μιλόσεβιτ και δεν σταμάτησαν με την εξαφάνιση του Μιλόσεβιτ. Συζητούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεχίζει το διάλογο. Αύριο συναντόμαστε με τον ε, κύριο Σανίνα που είναι ο νέο ηγέτη τη Γενική Διευθύνσεω και τον κύριο Χίτσλερ που είναι υπεύθυνο για το ΙΠΑ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξεπώνησε συνεδρίαση του Ζάγκρεπ το Μάιο, να συζητήσαμε το θέμα αυτό ένα έγγραφο τοποθέτησης που δείχνει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά στο θέσουμε ω εξή. Εξακολουθεί να είναι μετριοπαθέ. Εάν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο τολμηρή, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα το βουλγαρικό, έφυγε η κυρία Νεύσκη, να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Η Ευρώπη θέλει να έχει διασυνδέσεις βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά για το φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι ρωσικό το φυσικό αέριο παντού. Το θέμα του Ναμπούκο, του South Stream κλπ. Τα αφήνω στην άκρη για την ώρα. Ο Γκούτερ Oettinger ζήτησε από τον Υπουργό μας Ενεργείας και τον Ούγγρο Υπουργό Ενέργειας και μας είπε πρέπει εσείς παιδιά να φτιάξετε ε, μεταξύ Νης και Σόφιας να φτιάξετε αγωγό γιατί μετά θα έχουμε άλλη δίωδο για να εξισορροπήσουμε την παροχή φυσικού αερίου και αυτό είναι προς όφελος της Ευρώπης λόγω του όφελους του να είναι μέλος πήρε 65 εκατομμύρια ευρώ η, η Σόφια για ένα κομμάτι του αγωγού φυσικού αερίου που είναι έξι φορές πιο βραχής από αυτό που πρέπει να φτιάξει η Σερβία. Και ε, έχω, ε, στη Σερβία έχουμε πρόβλημα και έχουμε να περάσουμε και από ε, χαράδρα κλπ. Πρέπει να γίνει μελέτη ε, βιωσιμότητας τι θέλω να πω με όλα αυτά. Για 10 χρόνια τα καταφέραμε. Και δεν ήμουν πάντα στην κυβέρνηση. Να, τα, κατα... τα καταφέραμε αρκετά καλά. Έχουμε χαμηλό εθνικό χρέο. υγιές τραπεζικό σύστημα. Η μεγάλη Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει μόνοι μα να χρηματοδοτήσουμε όλα τα προγράμματα τα οποία ίσω και μπορώ να αποδείξω ότι 10 από αυτά τουλάχιστον έχουν μεγαλύτερο, ενδιαφέρουν περισσότερο την Ευρώπη από εμά. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μα. Δεν λέω ότι είναι άδικο διότι δεν πρόκειται να πετύχουμε κάτι έτσι, δεν έχουμε το οικονομικό, την οικονομική ισχύ, τη δυνατότητα να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Δεν λέω ότι πρέπει να τα κάνει η Ευρώπη αντί της ε, Σερβίας των Δυτικών Βαλκανίων. Λέω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να ωφεληθούν όλοι να ωφεληθούν και εκείνοι που συνεισφέρουν οικονομικά, διότι οι διαγωνισμοί θα, θα κερδιθούν από ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει καλέ δουλειέ, κυρίω για υποδομέ, για τι μεγάλε ευρωπαϊκέ εταιρείε, αλλά και τι μικρότερε ευρωπαϊκέ εταιρείε. Δεν σχολιάζω τι γίνεται με το, αυτά που κέρδισε η Πολωνία, ε, στην Πολωνία μάλλον που κέρδισαν ε, κινέζικε εταιρείε στο αυτοκινητοδρόμου. Ε, Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων. Τώρα, οικονομία αυτά που, μετά από αυτά που συνέβησαν στην Ευρωζώνη. Ξέρουμε ότι δεν θα μπούμε στην Ευρωζώνη για τουλάχιστον 20 χρόνια. Άρα το δινάριο θα είναι το νόμισμά μας. Αν έτσι έχουν τα πράγματα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε οικονομία με βάση το δινάριο και όχι με βάση το ευρώ. Διότι αν έχουμε με βάση το ευρώ την οικονομία ε, δεν θα έχουμε σωστή προσέγγιση. Θέλουμε βιώσιμο βιώσιμη θέση στον φάτη τρέχουσε συναλλαγέ. Άρα δεν πρέπει να παίζουμε με το χρήμα, να το αφήνουμε να ακολουθεί την πορεία του. Εν κατακλείδη, αυτό που κάναμε τα τελευταία τρία χρόνια. Πήγαμε στη Ουάσιγκτον και πήραμε τριετή διευθέτηση χωρίς να, να μας πιέζουν οι Βρυξέλλες ή το δούνου του. Διότι βλέπαμε το οικονομικό τσουνάμι να έρχεται, αυτό το κάναμε. Το κάναμε για να προσαρμοστούμε. Και εν γέννη ε, ήταν καλές οι επιδόσεις μας, αλλά οδήγησε στην ανεργία. Η ανεργία μας από 13,6 πήγε στο 19,6%. Η περιφερειακή, το όριο της φτώχειας πήγε από 6,2 στα 9,2. Και για τον κύριο Φάρου, λοιπόν, είμαστε σε καλά επίπεδα στον φάτσαν έχουν περιφερειακές διαφορές που πάνε από 1 μέχρι 7% από τις πλησιότερες γειτονιές του Βελιγραδίου μέχρι τις φτωχότερες περιοχές στα νότια και στα δυτικά και εκείνες οι περιοχές έχουν και αλβανι, αλβανικές μειονότητες, βοσνιακές μειονότητες οπότε είναι πιο σημαντική ε, η κάλυψη αυτών των διαφορών μόνο μερικά λεφτά απομένουν ε, τι να πω θα ήθελα να πω απευθυνόμενος προς εκείνο που έθεσε το ερώτημα το θέμα των ευρωσκεπτικιστών. Γιατί πρέπει να τα πληρώσει όλα αυτά η Γερμανία. Δεν πρέπει να τα πληρώσει η Γερμανία. Νομίζω ότι αυτό που συζητούμε ε, δεν είναι τα μεγάλα ποσά. Δεν τα ποσών είναι μεγάλα ή μικρά. Γνωρίζουμε πολύ καλά η ατμόσφαιρα οτι δεν είναι τέτοια που μπορούμε να ζητήσουμε να μας βοηθήσει η Ευρώπη. Το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό που προτείνουμε είναι να αναγνωριστούν καλύτερα τα προγράμματα εκείνα τα οποία είναι υποφελή για όλους. Να δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επικαιρό. Δεκέμβριος 2009 η Σερβία και αργότερα και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πέτυχαν την άρση των θεωρήσεων για τα ταξίδια. Τώρα 3,3 εκατομμύρια Σέρβοι πολίτες έχουν βιομετρικά διαβατήρια που κατασκευάζονται από βαβαρική τεχνολογία, με βαβαρική τεχνολογία την Μουλμπαουρ που ανοίγει εργοστάσιο στη Σερβία ε, για να ασχοληθεί με, τα, με διάφορα τα έγγραφα ασφαλεία. Και 6 εκατομμύρια των πολιτών μας διέσχισαν τα σύνορα Σέγγεν. Από τα 6 εκατομμύρια 17.000 είχαν πρόβλημα που ζήτησαν άσυλο. Αυτό ήταν αρκετό για να αλλάξει ο κανονισμός η νομοθεσία Σέγγεν. Αυτό ήταν αρκετό για να δημιουργήσει εντάσει μεταξύ τη χώρα μας της Σουηδίας, της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και του Βελγίου. Αυτό ήταν αρκετό για να γίνεται λόγος για ένταξη των Ρωμά. Εγώ είμαι πρόεδρος ε, του Συμβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου για την ένταξη των Ρωμά. Δεν είναι τυχαίο, είναι θέμα δεντολογικό, είναι θέμα ρεαλιστικής πολιτικής. 90% και αντί να μιλάω τεχνοκρατικά, να σας δώσω ένα παράδειγμα. 21 οικογένειες Ρωμά... στην μικρή πόλη Ποζάρεβατ. Και είναι αυτοί που τους διώξαν από το Κοσμοπέδιο. 200.000 Σέρβοι πολίτε είναι εσωτερικά εκτοπιστέντε από το Κοσμοπέδιο. Πολλοί από, αυτές είναι, από είναι Ρωμά. Αυτοί ζούσαν σε φρικτές συνθήκες. Φρικτές. Χάρη στο είπα... με 390.000 ευρώ καταφέραμε να φτιάξουμε 21 κατοικίες κατάλληλες για τους Ρωμά μόνο ε, με έναν όροφο, με κάποιους κοινόχρηστους χώρους κλπ. Γιατί είναι πολύ σημαντική κοινωνική ζωή για αυτούς. Πέρασε ένας χρόνος. Τέσσερις φορές το επισκέφτηκα ήδη. Γιατί τους είπα, θα ξαναγυρίσω, ε. Ποιοι είναι οι όροι για να εξακολουθούν να μένουν εκεί. Ότι όλα τα παιδιά τους θα πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Και όλα τα παιδιά τους πάνε στο σχολείο. Και ε, βάλαμε και βοηθούς για υποστήριξη, διότι δεν υπάρχει το αναγκαίο ανθρώπινο κεφάλαιο από την οικογένεια ως υποστήριξη. Ένα κοριτσάκι, ήταν 8 και χοροπηδούσε και μου έλεγε Είμαι χαρούμενη, είμαι χαρούμενη. Γιατί είσαι χαρούμενη, τη λέω, διότι τώρα μπορώ να μάθω. Τη λέω, δεν μπορούσε πριν. Λέει, Μα κύριε Τζέρι, δεν είχα ηλεκτρικό ρεύμα. Το χειμώνα λοιπόν δεν υπάρχει ήλιο, δεν υπάρχει φω, δεν υπάρχει μάθηση. Τα παιδιά λοιπόν πάνε στο σχολείο και η εμπειρία κατέδειξε ότι αυτή η παιδεία είναι ο καλύτερος τρόπος να θεδροποιηθεί ο κόσμος να ψάξει για δουλειά κλπ. Για, τι προσπαθώ να πω, ότι δεν ζητάμε από την Ευρώπη να κάνει τη δουλειά ημών, αλλά να εξετάσει προγράμματα κοινού συμφέροντο, όπου οι συνέπειες συνεργασία μπορεί να είναι υποφελεί για κοινωνικέ πτυχέ, για υποδομέ, για την ενέργεια, για την οικολογία, για τη γνώση. Και αν δείτε τα στοιχεία, δεν νομίζω ότι μπορεί να με πείσει κανείς ότι μόνο μία αναδιαρρύθμιση του συστήματος, διότι αυτό ζητούμε, θα κάνει τεράστια διαφορά. Μη λησμονείτε ότι βελτίωση στα Βαλκάνια επέτρεψε στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρώπη να μειώσει πάρα πολύ σημαντικά τον αριθμό των στρατευμάτων στο, στο Λοιπόν, πρέπει να μετήσει κανείς και τις, τις οικονομίες λόγω της ασφαλείας στα Βαλκάνια. Το κόστος που μειώθηκε τον, από τους ετούντες ε, άσυλο, από τους πρόσφυγες, ε, από τους εκτοπιστέντες. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση της ΕΦΤΑ που τα τελευταία χρόνια έδειξε ότι είναι μια διευθέτηση ε, εμπορική που αντιστάθηκε καλύτερα από οτιδήποτε άλλη περιοχή όσον αφορά το εμπόριο στην περιοχή μας. Και έχουμε σκεφτείτε το, συνεδριάς τακτικέ μεταξύ των Πρωθυπουργών, του Σέρβου, του Κροάτη και του Σλοβαίνου. Τι φορές έγινε τα, την, τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για προγράμματα. Η Σερβία, η Κροατία και η Σλοβενία δημιούργησαν μια εταιρεία Corridor 10 Freight. Freight διότι μπορούμε να ωφεληθούμε από τις υποδομές μας στον τομέα των μεταφορών των αγαθών τα επόμενα χρόνια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ξεκινάμε ήδη, ακόμα και αν αυτό ήταν ταμπού εδώ και 10 χρόνια, λέμε ότι ίσως αντί να έχουμε μικρές αεροπορικές εταιρείε που όλες χάνουν ε, χρήματα, να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Σκανδιναβοί με την ΣΑΣ ε, και με την ΤΖΑΤ παλιά, να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Σας είμαι θα γι' αυτό. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία. Δεν ζητάμε θαύματα δεν ζητήσαμε κάτι τέτοιο και δεν ζητάμε τον ουρανό μετάστρα. Δεν θέλουμε να ζητήσουμε τώρα τον ουρανό μετάστρα, αλλά με μικρή εμπειρία που έχουμε, δείτε με του μηχανισμού λειτουργήσαν αυτά που λειτουργήσαν, κοιτάξτε λίγο καλύτερα και τι συμφέρον κοινό έχουν τα Δυτικά Βαλκάνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το κάνουμε αυτό, ήδη κάναμε αρκετά, ούτω ώστε εμεί οι πολιτικοί, οι ντόπιοι πολιτικοί πρέπει να χειριστούμε τι προσδοκίε των πληθυσμών μα, που και αυτοί περνάνε την κρίση, να μπορέσουμε να έχουμε αρκετά εργαλεία στα χέρια μας για να κάνουμε να ζήσει η Ευρώπη στην περιφέρεια. Διότι αν δεν υπάρχει προσχώρηση, δεν υπάρχουν προγράμματα, δεν υπάρχουν σχέδια, σας ρωτώ, επί ποιες βάσεις μπορούμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα πρέπει τουλάχιστον ε, να ε, υπάρχει μια εικόνα, ένα ιδιώδες και ελπίζω και λίγη πραγματικότητα. Αυτά και ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρο που απαντήσετε σε όλες μας τις ερωτήσεις ομολογώ ότι εκείνοι μεταξύ ημών που πριν από 20 χρόνια με ματωμένη καρδιά είδανε η Ιουκοσλαβία να εκρήγνεται, να βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε ένα τμήμα η Σλοβενία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κροατία είναι στην διαδικασία διεύρυνση, η Σερβία βρίσκεται στη σωστή άγουσα και ακούγοντα τον δικό σα ενθουσιασμό, τη σαφήνεια, το δυναμισμό σα, μπορούμε να χαρούμε. Κατανοήσαμε το μήνυμα σα, ιδίω όσον αφορά την περίοδο που θα καλύπτω από το επόμενο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θα μεταβιβάσετε τι απόψει μα και οπωσδήποτε θα παραμείνουμε σε επαφή για να προσαρμόσουμε το διατακτικό το καλύτερο δικό. Ευχαριστώ. Πέρα συνεδρία.